και τα τοξικά απόβλητα. Όλοι γνωρίζουν τα αποτελέσματα της συνέπειας μιας κακής εξόριξης ε, πετρελαίου που μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στις κοινωνίες της γειτονικέ. Να μην ξεχνάμε πως φτάνουν οι παλιές τηλεοράσεις και οι παλιοί υπολογιστές στην Αφρική για να ανακυκλωθούν υποτίθεται, αλλά στην ουσία τα εγκαταλείπουμε σε μεγάλες χωματερές όπου εργαζόμενοι και πάρα πολλά παιδιά αναζητούν το χαλκό και το αλουμίνιο πριν τα κάψουν χωρίς καμία προστασία. Υπάρχει όμως και ένας θετικός δεσμός ανάμεσα στο περιβάλλον και την ανάπτυξη. Υπάρχει ένας τρόπος συνεισφορά στην οικονομική ανάπτυξη και την ανάπτυξη γενικότερα, επενδύοντας τις υπηρεσίες τις οποίες μας παρέχει η πλουσιοπάροχα η φύση. Λοιπόν, Αυτά είναι τα συμπεράσματα στα οποία θα μπορούσε να καταλήξει η ακρόαση αυτή. Θα πρέπει να διατηρήσουμε τις οικολογικές υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται από τα οικοσυστήματα πριν είναι πολύ αργά. Πριν το τίμημα το οποίο θα πληρώσουμε για την αποκατάσταση και διατήρηση των υπηρεσιών αυτών είναι πάρα πολύ ψηλό για να το δώσουμε. Σαν Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης θα ήθελα να καλωσορίσω τους εμπειρογνώμονες οι οποίοι σίγουρα θα συνεισφέρουν να είναι ενδιαφέρουσα η ακρόαση αυτή και να επιτρέψει να γίνουν ειλικρινείς και επικοδομητικές συζητήσεις. Τις ευχαριστώ και τους ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή τους και τους εύχομαι κάθε επιτυχία. Τώρα θα ήθελα να προσκαλέσω τους δύο συνυπευθύνους της ακροάσεως αυτής, την κυρία Λεύιν και την κυρία Τσίμα να πάρουν τον λόγο πλέον και να προεδρεύσουν στην ε, επόμενη φάση της ακρόασης. Κυρία Λόβιν, έχετε το λόγο. Ε, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλημέρα και καλώς ήρθατε όλοι στη συνεδρίαση αυτή για την ε, υποβάθμιση του περιβάλλοντος και θα ήθελα να πω ότι αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση που μπορώ να προεδρεύσω εγώ στο κομμάτι αυτό της ακρόασης για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και τη φτώχεια. Γιατί πολύ συχνά η υποβάθμιση του περιβάλλοντος για ορισμένους οδηγεί ε, σε περισσότερο πλούτο. Αλλά αυτό ισχύει μόνο για τους πλούσιους του κόσμου. Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος είναι αυτή η οποία έχει εξασφαλίσει την παραγωγή των φθηνών προϊόντων των, των οποίων όλοι χαίρομαι στη Δύση προς όφελος των πλουσιών όπως έλεγα αλλά ε, από παραγωγή των φτωχών. Παρατηρήσει λοιπόν ε, προκαταρκτικές. Καταρχάς ότι θα χρειαστεί δυστυχώς να αποχωρήσω νωρίτερα από ό,τι είχα προβλέψει. Όταν μου δοθεί το σύνθημα θα πρέπει να φύγω για την Επιτροπή Αλίας, όπου έχω ένα πολύ σημαντικό θέμα. Για την Αλία, πάλι σχετικό με τα ε, συστήματα και οι υπηρεσίες οικοσυστημάτων που χάνουμε. Ε, μια δεύτερη ανακοίνωση είναι ότι ο κύριος Ράσμουσεν από τη Δανία, ο οποίος επρόκειτο να παρουσιάσει μια ε, πρακτική μελέτη των συνεπειών <clears throat> της ανακύκλωσης αποβλήτων στην, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αναπτυσσόμενες χώρες. Δυστυχώς χτες μόλις μας ότι δεν μπορέσει να συμμετάσχει στην ακρόαση και δεν μπορέσαμε μέσα στην ε, την τελευταία στιγμή να ε, βρούμε αντικαταστάτη. Και έτσι αντί για αυτή την ε, παρουσίαση πρακτικού θέματος θα πρέπει να καταλήξουμε στη διατύπωση των συμπερασμάτων. Ε, εν τω μεταξύ όμως καλωσορίζω την κυρία Κέμπη, η οποία είναι επικεφαλής για την πρωτοβουλία για την περιβαλλοντική πολιτική προσανατολισμούς ε, του Ευρωπαϊκού ε, του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών στο Ναϊρόβι. έχει εργαστεί ως ε, σύμβουλος για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών. Ήταν εκπρόσωπος του ΙΣΥΠΑ της Αρμοστού για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, πάλι στο θέμα του περιβάλλοντος στην περιοχή των Μεγάλων στην υποστήριξη της διάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του Συμφώνου των Μεγάλων και για την προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των ε, κρατών της περιοχής με ειδικότητα προσέγγιση της ε, ανάπτυξης ανατολισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα. Πριν δώσω το λόγο στην Ιζαμπελ, η οποία θα κάνει την παρουσίαση για τα τελικά συμπεράσματα και τις συστάσεις του της αξιολόγησης ε, οικοσυστήματος για την ε, χιλιετηρίδα θα ήθελα να αναφερθώ πολύ σύντομα στα θαλάσσια οικοσυστήματα που υποβαθμίζονται ταχύτατα και που με ενδιαφέρουν εμένα ιδιαίτερα καθώς είμαι ενεργό και στην Επιτροπή Αλίας από την Επιτροπή Αξιολόγησης Οικοσυστημάτων καταγράφεται ότι πολλές από τις υπηρεσίες των οικοσυστημάτων ε, ε, υποβαθμίζονται με αποτέλεσμα να επιδεινώνεται η κατάσταση και ως προς τις στόχους της χιλιατηρίδας για την, προαγωγή, για την αντιμετώπιση μάλλον της φτώχειας και της πείνας. Το βλέπουμε αυτό ιδιαίτερα στα θελάσσια συστήματα, ότι δηλαδή 85% των ε, αλλιευμάτων ανά τον κόσμο είτε έχουν υπεραλλευθεί είτε έχουν προχωρήσει σε εξάντληση σχεδόν. Και αυτό το βλέπουμε όχι μόνο ε, ως προς τη σημασία του ε, ηχθείως ως ε, διατροφικού στοιχείου, αλλά και ως στοιχείο διαφύλαξης και προστασίας του θαλάσσιου οικοσυστήματος, αλλά και σε οικονομικούς όρους. Έχουν άλλωστε και η FAO και η Παγκόσμια Τράπεζα κάνει ανακοίνωση που γραμμίζουν τη σημασία για ολόκληρη την ανθρωπότητα των αλλιευμάτων η οποία δείχνει ότι χάνονται 50 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο λόγω της κακής διαχείρισης θαλάσσιων αλλιευμάτων. 3-3 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε 10 χρόνια εν ολίγης. Χάνουμε πολλά λοιπόν και σε οικονομικού όρου από την υπεραλίευση, από την εξάντληση των ελευθερικών επιθεμάτων Και τώρα, αν μου επιτρέψει, αγαπητοί φίλοι, θα θέλω να σα το λόγο για να μα κάνει την παρουσίαση για την ε, ε, αξιολόγηση της χειρετηρίδας. Ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Κέμφ. Ευχαριστώ πολύ, Ζαμπέλα. Είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε επιτέλους για την αντίληψη αυτή ότι η περιβαλλοντική προστασία και η ανάπτυξη είναι, αν... είναι αντικρουόμενοι όροι, όχι των αντίων. είναι όροι συμπληρωματικοί μεταξύ τους και είναι ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε προς μείωση των, ε, της ζημιάς του περιβάλλον ε, με παράλληλη την προσπάθεια για την ανάπτυξη. Θα ήθελα ξεκινώντας να καλωσορίσω και να καλημερίσω όλους τους φίλους και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τα θεσμικά όργανα, τα κόμματα, τα πολιτικά που βρίσκονται εδώ. Από τη UNEP, το Γραφείο των Βρυξελών, που είναι επίσης στη διαθεσή σας για συζήτηση μετά την παρουσίασή μας. Και σύντομα επιτρέψτε μου να αναφερθώ στην ε, αξιολόγηση οικοσυστημάτων της χιλιετηρίδας, τι σημαίνει, τι αφορά, πώς αναπτύσσεται, τι συνέπειες μπορεί να έχει, τι συνέχεια μπορεί να της δοθεί, φτώχεια και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες, ένα κοινό ε, πρόγραμμα του προγράμματος για την ανάπτυξη των Εθνών και της UNEP μαζί με τη Γενική Διευθύνση για την Ανάπτυξη και υποεθνική τεχνικές ε, αξιολογήσεις, δηλαδή μέσα στο, στην αξιολόγηση για τη χιλιατηρίδα, εθνικές ε, επιμέρους αξιολογήσεις ε, για δύο χώρες, τη Ρουάντα και την Ταϊλάνδη. Ξεκινώ αναφερόμενοι στο πλαίσιο για την αξιολόγηση της θα δείτε στις ε, υπηρεσίες ε, οικοσυστημάτων ότι αποτελούν βέβαια τα οικοσυστήματα τη βάση για την ανάπτυξή μας. Από αυτά αντλούμε τροφή αλλά και άλλα στοιχεία της εφημερίας μας όπως αναψυχή, καθαρά νερά, λίμνες, ε, ποτάμια, θάλασσες και επίσης μπορούν να αποτελέσουν και στοιχεία της έμεσες ε, έμεσες υπηρεσίες ε, που μπορούν να προσφέρουν τα οικοσυστήματα όπως αλλαγή στη χρήση των γεών, ειδική ε, εισαγωγή μάλλον ειδών, προσαρμογή τεχνολογίας, θεσμικό πλαίσιο, επιστήμη και τεχνολογία που μας λέει πώς μπορεί να γίνεται η διαχείριση του περιβάλλοντος και βέβαια πολιτιστικούς ή θρησκευτικού τρόπους διαφύλαξης ή συσχετισμού δια, ε, αλληλεπίδρασης το περιβάλλον και υπάρχουν και οι απευθείας ε, φορείς της αλλαγή όπως οι στη της όπως η εισαγωγή ε, η απάλληψη ειδών, προσαρμογή της τεχνολογίας, ε, κατανάλωση πόρων, εξωτερικές επεμβάσεις όπως φερειπίν αποξήρανση, όπως σε παραδείγμα άρδευση, όπως σε παραδείγμα την των δασών, κλιματικές αλλαγές στη συνέχεια ή άλλες ε, φυσικές, φυσιολογικές και βιολογικές ε, πρακτικές που επηρεάζουν, όπω είπα, όχι μόνο το περιβάλλον, το οικοσύστημα, αλλά και την ευημερία του ανθρώπου. Ερώτηση για το πώς μπορούν αυτοί οι φορείς να αλλάξουν τις υπηρεσίες του οικοσυστήματος και μέσω αυτού να επηρεάσουν την ευημερία του ανθρώπου και το επίπεδο του, το οικονομικό δηλαδή να οδηγήσουν στη φτώχεια. Ω προ την δημόσια υγεία αυτή επηρεάζεται βέβαια και από το περιβάλλον και από την ρήπανση, από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Η σχέση μας με το περιβάλλον αλλάζει. Παλαιότερα είχαμε σχέση περισσότερο με το υγιή και με το ε, δάσος και αυτό εκφραζόταν και στις διαπροσωπικές σχέσεις. Και αντίστοιχα και η ασφάλεια του ανθρώπου, η ελευθερία τη επιλογή, η δράση του ατόμου μέσα στην κοινωνία. Σημαντικό είναι εδώ λοιπόν να επισημάνουμε ότι οι υπηρεσίες οικοσυστημάτων όχι μόνο προσφέρουν ε, ε, τρόφιμα, καύσιμα και λοιπούς ε, πόρους για κατανάλωση του ανθρώπου, αλλά αποτελούν τμήμα της ζωής μας και χώρο μέσα στον οποίο εκφράζονται και πάνω στον οποίο στηρίζονται οι ανθρώπινες σχέσεις. Εν τέλει, όταν άρχισε η αξιολόγηση, όλη η συζήτηση που είχε να κάνει με το τι είναι οι υπηρεσίες οικοσυστήματος μας απασχόλησε και πάλι οι ε, κοινωνικές επιστήμες αλλά και οι φυσικές επιστήμες ε, στο βαθμό που ενεπλάκησαν με τους εκπροσώπους τους στην μελέτη αυτή ε, είπαν ότι πρόκειται για ένα ολιστικό σύστημα όχι μόνο δηλαδή τρόφιμα, νερό ή καύσιμα αλλά ταυτόχρονα και στήριξη του ε, κυκλικής κίνησης και της ανακύκλωσης του φυσιολογικού κύκλου δηλαδή την ε, διασφάλιση των εδαφών, την παραγωγή, τη δασική, τα είδη, τα θαλάσσια, τα θαλάσσια ε, οικοσυστήματα, το υγρό στοιχείο. Ταυτόχρονα όμως και επιδρούν το ένα πάνω στο άλλο αλλαγές κλιματικές, πλημμύρες και το καθεξής. Άρα έχουν πολύ σημαντική λειτουργία όλα αυτά τα συστήματα και όχι μόνο λειτουργία παραγωγής τροφίμων και νερού. Η πολιτιστική διάσταση είναι πολύ σημαντική. Επίσης, όπως είπα και νωρίτερα, Πολλοί, φαντάζομαι βγαίνετε εκδρομή το Σαββατοκύριακο, φεύγετε από τι Βρυξέλλες, ε, πάτε σε ένα δάσο ή μπορεί να πάτε μέχρι τη θάλασσα για το Σαββατοκύριακο. Είναι αυτή η διάσταση της αναψυχής και ανάπαυσης που προσφέρει η φύση το οικοσύστημα και πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση της, ε, των υπηρεσιών που προσφέρει το οικοσύστημα. το πού έλαβαν ε, χώρα και πότε. Μεταξύ του 2000 και του 2005 έγινε αξιολόγηση. 1.300 και άνω επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Είχαμε μια διεπιστημονική προσέγγιση και από τις κοινωνικές επιστήμες και από τις φυσικές επιστήμες στη μελέτη αυτή και αυτό που προσπάθησαν να κάνουν αυτοί οι επιστήμονες ήταν να καταγράψουν αλλαγές στο οικοσύστημα σύντο και οι αλλαγέ αυτές να δουν σε ποιο βαθμό έχουν επηρεάσει την ευημερία του ανθρώπου, την κατάσταση προ προς τη φτώχεια στις χώρες ή τι περιφέρειες που μελετήθηκαν και να προσφέρουν ε, διαφορετικές ε, προβλέψεις με τη μορφή σενάριου για το μέλλον. Η κλιματική αλλαγή φυσικά έχει πολύ μεγάλη σημασία στην προκειμένη περίπτωση και άρα προσπάθησαν να δώσουν διαφορετικές μεταβλητές ε, προβλέψεις ως προς το τι θα συνέβαινε αν έμενε η ίδια η χρήση γης, η ανάλαζε και τα λοιπά, η κατανάλωση, όλα αυτά για να δούμε σε ποιο βαθμό θα επηρεάζονταν το οικοσύστημα. Και αυτά μέσα στη συζήτηση για την ανάπτυξη και τη σημασία του περιβάλλοντος του οικοσυστήματος για την ανάπτυξη. Η αξιολόγηση αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί. Κάποια στοιχεία τα βλέπετε ήδη στις ε, ε, φωτοτυπίες. Έχουμε τα, τις διάφορες αξιολογήσεις ε, που έχουν ολοκληρωθεί που συνεχίζονται ακόμη ανά τον κόσμο. Κάποιες είναι περιφερειακές, κάποιες είναι εθνικές, κάποιες ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί. Κάποιες είναι ολοκληρωμένες και... Βλέπετε ότι προσπαθούμε να καταγράψουμε και την αντίληψη στην κάθε περιοχή για το τι είναι ο κόσμος. Στο Περού, Φερρυπίν, είχε συμμετοχή η κοινότητα Κιτσουά στις μελέτες μας ε, για να δούμε πώς βλέπουν το περιβάλλον, το οικοσύστημα και την ε, ευημερία. Τα έχουμε ενσωματώσει αυτά μέσα στις μελέτες μας. Τι συνέχεια δίνουμε στη μελέτη αυτή. Στόχος μου είναι ακριβώς να προσδιοριστεί ως αποτέλεσμα αυτής της μελέτης ε, ο τρόπος με τον οποίο θα χαράξουμε πολιτική, επαφάσεις που θα λάβουμε πολιτικές. Αξιολόγηση λοιπόν τι, σε τι βαθμό επηρεάζεται η εφημερία του ανθρώπου, τα διάφορα σενάρια ανά τον κόσμο. Από εδώ και μπρος λοιπόν τι θα κάνουμε, πώς πραγματικά επηρεάζεται ο αρμόδιος να λάβει αποφάσεις, εάν επηρεάζεται, ποιος είναι αυτός ο αρμόδιος, και πώς τα επιστημονικά αυτά στοιχεία μπορούν να είναι χρήσιμα για τη χάραξη πολιτικής. Το πρώτο πράγμα που κάναμε στο follow-up ήταν να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο για την ανάπτυξη ε, δυνατοτήτων ε, στις διάφορες χώρες μεταξύ αυτών που το ήθελαν, που το επιθυμούσαν, ανταλλαγή εμπειριών για τις διάφορες ε, μελέτες και με βάση τις εμπειρίες και τα διδάγματα που αποκομίσαμε ε, οικοδομήσαμε προτάσεις για την παγκόσμια ατζέντα και τον διάλογο. Η διακυβερνητική πλατφόρμα για την ε, διαχείριση των οικοσυστημάτων και τη διοπικιλότητα που βλέπετε εδώ είναι ένα διακυβερνητικό σώμα που αξιοποιεί την μελέτη αυτή για να ενημερώνει τους ε, πολιτικούς, ε, τους αρμόδιους για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων. Πέραν αυτού, αναπτύχθαμε και ένα εγχειρίδιο που εξηγούμε την μεθοδολογία μα, τα διάφορα σενάρια που έχουν αξιοποιηθεί, τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να κάνει κανεί τη δική του εκτίμηση στη χώρα του, στην περιοχή του, στην περιφέρειά του, τα διάφορα εργαλεία μπορεί να κανεί να αξιοποιήσει. bit about the Poverty Environmental Initiative. Um, as I said before, this is UNDP UNEP uh, initiative. Προσπαθούμε λοιπόν με τη μελέτη αυτή που αναπτύσσεται στα πλαίσια του προγράμματος για την ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών να στηρίξουμε σε εθνικό και υποεθνικό και εσωτερικό δηλαδή πρόγραμμα, επίπεδο, προγράμματα, κυρίως για αναπτυσσόμενες χώρες, 18 τον αριθμό αυτή τη στιγμή, στην ανάπτυξη ε, προγραμμάτων για την ε, βελτίωση σύνθεσης ε, και της σχέσης περιβάλλοντος και ανθρώπων. Κυρίως με τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών Προγραμματισμού Ανάπτυξης αλλά και, την, το πρόγραμμα για την ανάπτυξη των Εθνών. Δηλαδή, Βοηθούμε και τη χώρα και τα Ηνωμένα Έθνη να αναπτύξουν ε, διαλειτουργικούς δεσμούς μεν, αλλά ταυτόχρονα και να βρεθούν οι πόροι από τους εθνικούς προϋπολογισμούς ώστε να αξιοποιηθούν σε πολιτικές που θα ωφελούν τους φτωχούς παράλληλα με το περιβάλλον. Στα διδάγματα που έχουμε αποκομίσει απευθυνόμενοι σε χώρες όπως η Τανζανία και η Ουγκάντα έχουμε εξηγήσει τα προγράμματά μας. Τα προγράμματα δηλαδή πρέπει να έχουν σωστά σημεία εισόδου ή εκκίνησης και υπογραμμίζω σε επίπεδο εθνικό εμείς από το UNDP δεν μιλάμε με ε, Υπουργεία Περιβάλλοντος αλλά με Υπουργεία Οικονομικών οικονομικών προγραμματισμού και ανάπτυξης και προσπαθούμε στους αρμόδιους φορείς να εξηγούμε τι είναι σημαντικό, ποιος είναι ο σύνδεσμος μεταξύ οικοσυστήματος και μείωσης της φτώχειας. Προσπαθούμε να κάνουμε τις αξιολογήσεις μας από κοινού, μαζί τους, σε συνεργασία μαζί τους δηλαδή. Και επίσης πολύ σημαντική είναι η οικονομική ανάλυση εναλλακτικών χρηστών οικοσυστημάτων. Τα οικονομικά επιχειρήματα είναι εκείνα τα οποία είναι πιο γρήγορα και πιο εύληπτα κατανοητά, οικονομικά δηλαδή, απευθυνόμενα στα οικονομικά υπουργεία, που αντιλαμβάνονται πιο εύκολα όταν του εξηγούμε σε οικονομικού όρου ποια είναι η χρησιμότητα του οικοσυστήματο και πώ μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση τη φτώχεια. Ταυτόχρονα, ωστόσο, προχωρούμε και περισσότερο <clears throat> ώστε να εξασφαλίσουμε εμπλοκή ε, άλλων παραγόντων ε, και εταίρων όπως πέραν των βουλευτών ε, που βεβαίως πρέπει να παρακολουθούν τις αποφάσεις σχετικά με τις δημόσιες δαπάνες, επενδύσεις, ξένες επενδύσεις, αξιολόγηση. Τους μαθαίνουμε να χρησιμοποιούν την αξιολόγηση περιβάλλοντος ή οικοσυστήματος ώστε να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις, να παρακολουθούν την τήρηση των ε, αποφάσεων και βέβαια να έχουν επιλογές εναλλακτικέ πολιτικές. Μαζί με αυτούς όμως απευθυνόμαστε και σε κοινωνικούς εταίρους όπως Γεωργοί και άλλοι και απευθυνόμαστε και σε λύσεις, στρεφόμαστε και προς λύσεις ανάπτυξης νοτήτων για να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές πιο συγκεκριμένα. Επανέρχομαι μάλιστα τώρα από το ΛΑΟΣ, όπου το Εθνικό Ερευνητικό Ινστιτούτο Συνεργασία με το Εθνικό Υπουργείο Ανάπτυξης προέβη στη δική του αξιολόγηση οικοσυστήματος, αναζητώντας τις επιπτώσεις των μέσων αλλοδαπών επενδύσεων στα οικοσυστήματα από την παραδοσιακή ε, ορίζοκαλλιέργεια έχουν περάσει ε, στο καουτσούκ και σε άλλες καλλιέργειες και θέλουν να μελετήσουν πώς άλλαξαν οι συνθήκες εργασίας, παραγωγής, διαβίωσης των ε, στις διάφορες περιοχές, πώς επηρεάστηκαν διάφορα στρώματα της κοινωνίας από την εξέλιξη αυτή και νομίζω ότι από την ε, ανάλυση αυτή βλέπουν όχι μόνο πόσο άλλαξαν οι υπηρεσίες οικοσυστημάτων αλλά και η κατάσταση σε σχέση με τη φτώχεια, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο ο κόσμος βλέπει τη γη και νομίζω τους ε, δείξαμε ότι είναι πολύ σημαντική η οικονομική ανάλυση. Ε, ταυτόχρονα όμως συνειδητοποιούν ότι για τον κόσμο σημαντική είναι όχι μόνο η οικονομική διάσταση του εισοδήματο, αλλά και η ασφάλεια και η ευημερία και η πρόσβαση σε καθαρά νερά, όχι δηλαδή μολυσμένα και η δυνατότητα να ζουν μαζί με την οικογένειά τους, η δυνατότητα να σχεδιάζουν το μέλλον ε, μαζί με τα παιδιά τους. Όλα αυτά τα στοιχεία δηλαδή φαίνονται πολύ σημαντικά και επιτρέπουν ε, να καθοδηγήσουμε τη λήψη των αποφάσεων ως προς το μέλλον, ε, της απευθείας ξένες επενδύσεις, την χρήση της γης και την ε, κατεύθυνση που θα πάρουν οι επενδύσεις. Όλα αυτά τα ενδιαφέροντα πολύ και το Κοινοβούλιο του λαού ανέλαβε πολύ ενδιαφέροντα ρόλο. πολύ ενεργό ρόλο στην υπόθεση αυτή. Ήταν πολύ ενδιαφέρον και θα είναι πιστεύω ενδιαφέρον αν επιτροπές όπως η δική σας μπορούσαν να τους ε, δώσουν, ε, να τους προσφέρουν την εμπειρία τους ε, για τις επενδύσεις αυτές, για το περιβάλλον και τις υπηρεσίες οικοσυστήματος. Επίσης αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε κυβερνήσεις που μπορεί να μας δώσουν κάποιες ενδείξεις για την αξιολόγηση και την επιτήρηση και προσπαθούμε το mainstream, ε, η εισαγωγή δηλαδή της διάστασης της φτώχειας στο περιβάλλον να γίνεται κατά τρόπον ώστε οι πιστώσεις ε, από τον προϋπολογισμό να στρέφονται περισσότερο προς ε, πολιτικές για την αντιμετώπιση της φτώχειας και την πρόσκληση του περιβάλλοντος και μαζί με την ανάπτυξη θεσμικών δυνατοτήτων και υποδομών να ενισχύουμε το περιβάλλον. Αυτό βέβαια έχει να κάνει και με την ε, έρευνα. Πρέπει να πούμε ότι στο Λάος η κυβέρνηση ήταν διατεθειμένη να ακούσει τις συστάσεις του Ερευνητικού Ινστιτούτου. Ε, όμως για μας ήταν η πρώτη φορά και η ο προβληματισμός μας ήταν πώς θα μπορούσαμε παράγοντες της οικονομίας και της κοινωνίας όπως ε, συνδικαλιστικά σωματεία, γεωργούς, μη κυβερνητικέ οργανώσεις να τους φέρουμε σε, μέσα στη συζήτηση αυτή και την αντιπαράθεση απόψεων και πώς θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν το πρόγραμμά μας να το οικοδομήσουμε κατά τρόπο χρήσιμο και πιστικό ώστε οι συζητήσει να μην περιοριστούν μόνο σε δημόσιε διαβουλεύσει, αλλά να οδηγήσουν μια πραγματική ανταλλαγή απόψεων. Γιατί ορισμένε μη κυβερνητικέ οργανώσει με είχαν ερωτήσει τι ακριβώ ε, προβλέπουμε και πώ μπορούμε να προσδιορίσουμε για το μέλλον τι επαφέ αυτέ, αν θα ήταν απλώ συμβουλευτικέ, μόνιμε συμβουλευτικέ επαφέ ή κάτι άλλο. Συνοπτικά τώρα η προσέγγιση. Έχει σημασία βέβαια να είμαστε παρόντες στον προσδιορίζεται η, η ατζέντα προγραμματισμός δηλαδή για το περιβάλλον κατά της φτώχειας, κοινωνικά, οικονομικά κριτήρια και επιχειρήματα με την αξιολόγηση που έχουμε κάνει, γιατί γίνεται αυτό, γιατί ε, λαμβάνονται συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές με, τις τεχνικές, με τεχνική υποστήριξη, με την δυνατότητα αξιολόγησης και εκτίμησης των συνεπειών της χάραξης πολιτικής και την εμπλοκή όχι μόνο κυβερνητικών φορέων ή κρατικών αλλά και μη κρατικών φορέων. Όπως είδατε επίση χρησιμοποιούμε ε, για τα δικά μας προγράμματα την αξιολόγηση οικοσυστήματος για να δείξουμε στους ε, ε, φορείς του αρμόδιου για τη λήψη των αποφάσεων, πόσο μεγάλη σημασία έχουν, ε, πόσο μεγάλη σημασία έχει η συμμετοχή των παραγόντων της κοινωνίας, μη κυβερνητικών οργανώσεων, γεωκτημόνων και το καθεξής και ήθελα να εξηγήσω επίσης και για τα, με τα δύο παραδείγματα της Θελάντης και της Ρουάντα πόσο επηρεάστηκε και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων και πόσο σε μακροχρόνιο επίπεδο μπορεί να επηρεαστεί η δυνατότητα και η βούληση για λήψη αποφάσεων και για χάραξη πολιτικής. Θα ήθελα επίσης να δώσω ένα μικρό πρόγραμμα θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε μια οικονομική ανάλυση του, διαχείριση της διαχείρισης φυσικών πόρων που έχει λάβει η χώρα στη Ρουάντα, όπου εξέτασαν και την περιοχή των Ελλών αλλά και των δασών και διαπιστώνουν ότι δύο σημαντικέ ε, πτυχές της υποβάθμισης είχαν να κάνουν με την δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Ξέρετε ότι η Ρουάντα έχει σχεδόν 100% υδροηλεκτρική ενέργεια. Επομένως, υποβάθμιση των ελών των, ε, του, του υγρού στοιχείου αλλά και των δασών έχει οδηγήσει υποβάθμιση αυτής της ικανότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Έχουν αποξηρανθεί τα έλλη, έχουν κοπεί τα δάση, δεν υπάρχει σταθερή παραγωγή και προσφορά ε, ηλεκτρικού ρεύματο με σημαντικές διακοπές ρεύματο ε, που διαταράσσουν όλο τον ε, κοινωνικό και οικονομικό βίο. Ταυτόχρονα βέβαια μείωση και των εσόδων που διαπιστώνουν και οι αρμόδιοι για την πολιτική φορείς ότι υπάρχει σαφής διασύνδεση μεταξύ υποβάθμισης οικοσυστήματος και οικονομικής δραστηριότητας και δυνατότητας για βιομηχανική παραγωγή και αναλογίζονται τι θα πρέπει να κάνουν από εκεί και πέρα. Τι κάνουμε λοιπόν, η αξιολόγηση οδηγεί σε πολιτικές για τη μείωση της φτώχειας που είχαν από κοινού με την Παγκόσμια Τράπεζα στις οποίες πλέον βλέπουν και τη διάσταση του περιβάλλοντος όπως είπα, σημαντική διάσταση της ε, μείωση της παραγωγής της ροπητικής ενέργειας στην οικονομία και αυτό που μπορούσαμε να συζητήσουμε λοιπόν μαζί τους ήταν να πούμε ωραία τι μπορούμε να κάνουμε, ολοκληρωμένο προγραμματισμό, ενημέρωση ε, μεταξύ Υπουργείων ε, ενέργειας, προγραμματισμού δημόσιας υγείας, δημόσια διαβούλευση, καθώς η Ρουάντα δεν έχει μόνο την ετήσια εθνική διαβούλευση που γίνεται το Δεκέμβριο, αλλά είχε και από επίπεδο επαρχίας και από επίπεδο ε, νομού αναπτύξει συζητήσεις σε ομάδες με θέμα το τι συμβαίνει, ποια είναι τα πρακτικά βήματα και ποιο μπορεί να είναι το πρόγραμμα για την ανάπτυξη και την βοήθεια προς τους φτωχούς. Επομένως, Έγινε όλη αυτή η συζήτηση για το γεγονός ότι η υποβάθμιση του οικοσυστήματος συνδέεται ε, με το εισόδημα από την υδροηλεκτρική ενέργεια και γίνεται εθνική συζήτηση στη χώρα αυτή. Και γι' αυτό έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αποκατάστασης του υγροβιότοπου αυτού και γίνεται εκτελείστε αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο πρόγραμμα αναδάσωσης ώστε να βοηθηθεί ο πληθυσμός να δημιουργηθεί εισόδημα για τους ε, κατοίκους εκεί και να έχουμε νέες εγκαταστάσεις, σταθμούς υδροελεκτρικής ενέργειας έτσι ώστε να προχωρήσει η ανάπτυξη. Στην Ταϊλάνδη τώρα. Η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης ζήτησε να γίνει αξιολόγηση των οικοσυστημάτων σε τρεις επαρχίες και βασική ιδέα εδώ ήταν να ε, υπάρχει καλύτερη ενημέρωση για τον εθνικό σχεδιασμό βασικό ερώτημα είναι το εξής. Πώς μπορούμε να έχουμε αναπτυξιακές πολιτικές οι οποίες να περιλαμβάνουν και την ανάπτυξη της γεωργικής δραστηριότητας ενώ παράλληλα ε, να περιλαμβάνουν και τις προσπάθειες διατήρησης των οικοσυστημάτων να δημιουργηθούν εισοδήματα και να υπάρχουν προγράμματα καταπολέμησης της φτώχειας. Όπως θα δείτε σε αυτές τις τρεις διαφάνειες, οι αλλαγές χρήσης γης με την αποψήλωση των δασών. Μεταξύ άλλων, από το 1977 μέχρι το 2009 έχουν, είναι εξελίξεις που έχουν επηρεάσει πολύ αρνητικά τα οικοσυστήματα. Η συζήτηση ήταν αρκετά συμμετοχική και έτσι η ίδια η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης αποφάσισε να προσφέρει χρήματα για να γίνει περαιτέρω διαβούλευση με τους διαφόρους εμπλεκόμενους φορείς στις διάφορες περιφέρειες, προκειμένου να καταρτιστούν διάφορα σενάρια για εναλλακτικέ χρήσεις γης για τις συγκεκριμένες τρεις επαρχίες. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο λειτουργούμε, πώς συνεργοζόμαστε με τις διάφορες κυβερνήσεις στις διάφορες περιοχές. Βεβαίως ε, είμαστε ευγνώμονες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία μας προσφέρει μεγάλη στήριξη. Ε, είναι διαφορετικού είδους ε, εταίροι και δωρητές οι συνομιλητές μας. Ο συνάδελφος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω ότι θα πάρει τώρα το λόγο και θα μας πει η συνάδελφος πώς υποστηρίζει αυτού του είδους τις πρωτοβουλίες, πώς μπορεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μας βοηθήσει πώς μπορείτε να αξιολογήσετε αυτές τις αξιολογίες να χρησιμοποιήσετε αυτές τις αξιολογήσεις. Ε, αυτά προς το παρόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, uh, Isabel Kempf. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, λέει η Πρόεδρος, για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας. Θα δώσω τώρα το λόγο στους συναδέλφους να σχολιάσουν ή να θέσουν ερωτήματα ενδεχομένως. Bob Keller. είναι η συνάδελφος που θα με αντικαταστήσει, θα προεδρεύσει και τη δίνω το λόγο για την πρώτη ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας, ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Νομίζω ότι αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μπορεί να αξιολογηθεί η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, αλλά να γίνει συνάμα και κάτι γι' αυτό το πρόβλημα. Μα είπατε πολλά για τη διαδικασία, για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται, για τον αντίκτυπό τη. Μπορείτε να μα πείτε και δύο λόγια για τα αποτελέσματα, τα συνολικά. Ε, διαφαίνονται συγκεκριμένες τάσεις ε, για συγκεκριμένε περιοχέ που έχουν πληγεί ιδιαιτέρω. Ε, θα ήταν ενδιαφέρον ε, αν υπάρχουν τέτοια στοιχεία διαθέσιμα. Ευχαριστώ. Να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Γκαρθία Διαστεμέρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την ε, Επιτροπή για την πρωτοβουλία που ανέλαβε. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω το εξής ε, ε, την ομιλήτρια. Ως προς το πρόγραμμα της Ρουάντα, λαμβάνουν υπόψη τους τον πόλεμο, τις συγκρούσεις μεταξύ των Χούτου και των Τούτσι ως στοιχεία καθοριστικά, οι συγκρούσεις εννοώ, για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Λαμβάνουν υπόψη τους τη σύνδεση μεταξύ περιβάλλοντος και φτώχειας με ε, τις συγκρούσεις μεταξύ Χούτου και Τούτσι. Ευχαριστώ πολύ. Mr. Cortés Lastra. Ο κύριος Κορτές τώρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ και εγώ με τη σειρά μου την ε, ομιλήτρια για τη συμμετοχή της σε αυτή τη δημόσια ακρόαση στη Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή, για την παρουσίασή της. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες που μας ε, έθεσε υπόψη. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποιους, προβληματιστι... κάποιους προβληματισμούς. Αυτή τη στιγμή ε, συμβαίνει στον κόσμο ακριβώς το αντίθετο από τον τίτλο της δημόσιας ακρόασης. Δηλαδή, η μείωση της φτώχειας έχει ένα τεράστιο περιβαλλοντικό κόστος. Μπορούμε να μιλήσουμε για τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία, την Κίνα, για παράδειγμα. Πάρα πολλά μέτρα αναπτυξιακά εφαρμόζονται οδηγούν στην ανάπτυξη και το τίμημα το περιβαλλοντικό που καταβάλλεται είναι τεράστιο. Είναι κάτι το οποίο γνωρίζουμε όλοι. Και βεβαίω γι' αυτό θα πρέπει να σα ευχαριστήσουμε για την προσπάθεια που καταβάλλετε να παρέχετε εναλλακτική λύση ε, εναλλακτικέ ιδέες για το πώς θα αναπτυχθούμε τελικά, για το πώς πρέπει μια χώρα να αναπτύσσεται και πώς πρέπει μια χώρα να λειτουργεί και να δουλεύει. Και ταυτοχρόνως μας προσφέρετε εναλλακτικέ λύσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα, πρέπει να λειτουργήσουμε για να πετύχουμε την εξάλληψη της φτώχειας που είναι και βασικός στόχος των εργασιών μας στην Επιτροπή μας. Έχω λοιπόν την εξής ερώτηση. Ε, την περίπτωση της Ρουάντας. Μας εξηγήσατε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το 100% ε, ε, ε, εξάρτηση από τους σταθμούς παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας, ε, προσπάθειες εμπλοκής και συμμετοχής του συνόλου της ε, κοινωνίας ε, σε αυτή τη συζήτηση για τη διαχείριση των ενεργειακών πόρων στη Ρουάντα και ούτω καθεξής. Και στο τέλος της παρουσίασής σας μας είπατε ότι θα έχουμε νέους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υδάτινους πόρους δεν υπάρχει αναλεκτική με το δεδομένο του βαθμού αποψήλωσης ε, ε, των δασών στη χώρα αυτή. Δεν είμαστε ικανοί, δεν μπορούμε να ενσωματώσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη χώρα αυτή, να μπορεί να είναι ένα ενδεχόμενο να αρχίσουμε να δουλεύουμε πάνω στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη χώρα αυτή, ώστε ίσως να αντικατασταθεί ε, να αντικατασταθούν οι υφιστάμενες πηγές ενέργειας από ανανεώσιμες σε βάθος χρόνου. Και, επίσης, ε, έχετε σκεφτεί ποια είναι η σχέση μεταξύ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξάλληψης της φτώχειας. Είναι κάτι που σας προβληματίζει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Σίμερ παρακαλώ. Και από πλευρά μου θα ήθελα να εκφράσω τι θερμέ μου για την συμμετοχή σα και την ομιλία σα και να ρωτήσω, όπω και ο νωρίτερα, την ε, επίδραση και της ανάπτυξης στην ε, καταστροφή του περιβάλλοντος, αλλά και αντίστροφα θα ρωτούσα εγώ, συγκεκριμένα κλιματική αλλαγή και καταστροφή του περιβάλλοντος και σχέση τους με την φτώχεια, την πείνα και βέβαια την καταστροφική κατάσταση στη Σομαλία που γνωρίζουμε φέτος. Από την εμπειρία που έχετε, μπορεί η πολιτικός υπεύθυνη στις χώρες αυτές αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο μέσα στην ΕΕ να αντιληφθούν ότι υπάρχει αυτή η αδιάρρηκτη σχέση μεταξύ περιβάλλοντος καταπολέμηση, δηλαδή κατά, καταπολέμηση της καταστροφής του περιβάλλοντος, ταυτόχρονα βαίνει και φέρνει αποτελέσματα και στην, στον αγώνα για την καταπολέμηση της φτώχειας. Ευχαριστώ κύριο Γκέρενς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι ένα από τα προβλήματα τα πιο σημαντικά έγκυται στο γεγονός ότι η δεν είναι προτεραιότητα για τις αναπτυσσόμενες χώρες η προστασία, η διατήρηση ε, των δασών. Και εξηγώ τι θέλω να πω. Έχουμε μια εταιρική σχέση, επομένως αφού κραζόμαστε τις ανάγκες των εταίρων μας από τις χώρες του Νότου. Και σε αυτό το πλαίσιο, ε, αν, αν μας προτείνονται σχέδια διατήρησης ε, των δασών, δεν υφίσταται απάντηση από τη δική μας πλευρά. Πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτή τη δυσκολία. Αναφέρομαι ε, σε ένα πρόγραμμα το οποίο είχα παρακολουθήσει εγώ προσωπικό στην Μπουρκίνα Φάσο. Ε, λίγα εκτάρια, λίγες εκατοντάδες εκτάρια απομένουν από ένα πολύ μεγάλο δάσος στη χώρα αυτή. Ήταν πρόβλημα να πιστεί ο πληθυσμός να ξαναφυτέψει δέντρα γύρω-γύρω από αυτό το δάσος. Προκειμένου να ε, έχει επαρκή ξυλία για τις ανάγκες των οικοκυριών. Και μόλις ε, πετύχαμε αυτή τη φύτευση, μπορέσαμε, θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε μέτρα για τη διατήρηση των ε, πόρων αυτών. Είναι ένα πρόγραμμα που ε, ε, εκτείνεται σε βάθος χρόνου 20 ετίας και απαιτεί φυσικά ισχυρή πολιτική βούληση από τις αρμόδιες εθνικές και τοπικές αρχές. Και πολύ συχνά μας, λέει, μας αναφέρεται ότι στην καταπολέμηση της φτώχειας οι προτεραιότητες πρέπει να είναι άλλες. Ερωτώ λοιπόν πώς μπορούμε να αυξήσουμε την συνειδητοποίηση, αν θέλετε, των πολιτικών ηθινόντων. Πώς μπορούμε να τους κάνουμε να ε, νιώσουν περισσότερο ε, την ανάγκη να προστατευτούν οι δασικοί πόροι. Τι χρειάζεται για να είμαστε περισσότερο πιστικοί. Καλώς. Πριν δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και εγώ έχω μια ερώτηση να σας υποβάλω. Ποιο είναι το βασικό εμπόδιο, κατά τη γνώμη σας, ε, ποιος είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων δεν λαμβάνεται τόσο πολύ υπόψη στη, κατά τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Η ε, κλειδί για την ε, λύση του προβλήματος είναι η ατζέντα Ρίο συν Πώς μπορούμε να συμβιβάσουμε τα βραχυπρόθεσμα οικονομικά ωφέλη ε, και να ε, μπορέσουμε να τα ε, συνδυάσουμε με την μη υποβάθμιση του περιβάλλοντος σε βάθος χρόνου. Να δώσω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον αναπληρωτή προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαχείριση των υδάτων και την προστασία του περιβάλλοντος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Όπως ακούσαμε, ένα από τα βασικά ευρήματα της αξιολόγησης των οικοσυστημάτων για τη χιλιετία είναι ότι η υποβάθμιση ε, των, του περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων είναι ένας από τους βασικούς λόγους μη επίτευξης των στόχων της χιλιετίας. Επομένως η σχέση είναι άρρηκτη και είναι προφανής. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε ε, γι' αυτό και στο πλαίσιο της αναπτυξιακής βοήθειας. Από τη στιγμή που στόχη της ε, αναπτυξιακής βοήθειας είναι η μείωση της φτώχειας, η επίτευξη των στόχων της εχιλιετίας και η προστασία του περιβάλλοντος. Νομίζω λοιπόν ότι δικαίως μπορούμε να πούμε ότι στο παρελθόν αλλά και σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέκαθεν ε, κρατούσε τα ενία ε, στον αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος και πάντοτε αυτό το έθετε στο προσκήνιο ακόμα και στις εξωτερικές της σχέσεις. Ε, εδώ και πολλά χρόνια έχουμε περιλάβει τη συνιστόσα του περιβάλλοντος σε όλων των ειδών της συνεργασίας μας, σε επίπεδο χάραξης πολιτικής, προγραμματισμού δράσεων και εφαρμογής και υλοποίησης των δράσεων. Θα ήθελα πρώτα να θίξω το θέμα ε, της χάραξης πολιτικής. Το 2005 είχαμε την Ευρωπαϊκή Συνένωση για την ανάπτυξη και εκεί δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια της αηφόρου ανάπτυξης και προβλέψαμε υποχρέωση μεταξύ άλλων ε, χρήσης αξιολόγησης περιβαλλοντικών αντικτύπων να γίνουν δηλαδή οι αξιολογήσεις και οι μελέτες αυτές τα εργαλεία για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε ε, την εικόνα που επικρατεί στις χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Έχουμε επίσης την ε, ατζέντα για την αλλαγή τη νέα περιβαλλοντική μας πολιτική. Και βασικό μας σλόγγαν εκεί είναι η βιώσιμη και συμπεριληπτική ε, αηφόρο ανάπτυξη, η χρηστή διακυβέρνηση και η δημοκρατία. Η ανάπτυξη βεβαίως δεν είναι αηφόρος εάν ε, πλήττει το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα και τους φυσικούς πόρους πάνω στους οποίους στηρίζεται. Γίνεται μνήα στην προώθηση της πράσινης οικονομίας και τονίζονται δύο βασικοί τομείς, αηφόρος γεωργία και αηφόρος ενέργεια. Στη συνέχεια το ερώτημα είναι πώς οι πολιτικές αυτές θα μεταφραστούν σε πράξεις. Και γι' αυτό έχουμε αναπτύξει εργαλεία, μεθοδολογία, την οποία έχουμε προσφέρει στους συναδέλφους μας, έτσι ώστε να μπορέσουν να ενσωματώσουν τα θέματα του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής σε όλα τα σχέδια και τα έργα που θα εφαρμόσουν και που θα κάνουν στη συνέχεια. Έχουμε λοιπόν καταρτήσει κατευθυντήριες γραμμές ε, έτσι ώστε το περιβάλλον και η κλιματολογική αλλαγή να ε, ε, είναι στο επίκεντρο κάθε πολιτικής και κάθε προγράμματος που εφαρμόζεται και έχουμε περιβαλλοντικά προφίλ αναχώρα τα οποία είναι ένα υποχρεωτικό εργαλείο πρέπει να υπάρχουν για κάθε χώρα αναπτυσσόμενοι και μη. Έχουμε την στρατηγική αξιολόγηση για το περιβάλλον, την αξιολόγηση περιβαλλοντικού αντικτύπου και την αξιολόγηση κινδύνων για το κλίμα. Βάσει των ε, χρηματοδοτικών μέσων έχουμε μια συγκεκριμένη θεματική γραμμή του προϋπολογισμού ε, που είναι αφιερωμένη στο περιβάλλον, αποκλειστικά και μόνο. 1,1 δις είναι ο προϋπολογισμός της ε, δημοσιονομικής αυτής γραμμής για το υπάρχον, το υφιστάμενο δημοσιονομικό πλαίσιο 2007 με 2013. Ε, με αυτά τα χρήματα ε, αναπτύσσονται, εφαρμόζονται προγράμματα στις αναπτυσσόμενες χώρες αναφορικά με τα χημικά, την ποιοποικιλότητα, την καταπολέμηση της αποψήλωσης των δασών μεταξύ άλλων. Και στηρίζουμε διάφορα έργα που έχουν να κάνουν με τα ηλεκτρονικά απόβλητα και στηρίζουμε και το πρόγραμμα που παρουσιάστηκε προλίγου. Ε, έχουμε προγράμματα για απαξιωμένα ζυζανιοκτώνα και έχουμε και τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κοπεχάγη ε, για την προστασία του κλίματος, για την ε, αηφόρο παραγωγή και μέρος των χρημάτων δίδονται για τις ε, διεθνείς συμφωνίες και για την εφαρμογή των προβλεπωμένων της ε, Σύμβασης για τη Βιοπικιλότητα, για την καταπολέμηση της απερίμωσης και της αλλαγής του κλίματος. Αυτές είναι οι βασικές παρατηρήσεις που είχα να κάνω ως προς τις ε, θεματικές ενότητες. Έχουμε και γεωγραφικά εργαλεία το Ίντρα ECP, βάση του EF. Έτσι, εκεί, σε αυτό το πλαίσιο, στηρίζουμε ε, την, ε, ε, στο πλαίσιο των διμερών συμφωνιών, στηρίζουμε την προσπάθεια για να υπάρξει αυτό το οποίο αποκαλούμε capacity building, απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων από πλευράς της αναπτυσσόμενης χώρας. Προσπαθήσαμε στις προγραμματικές κατευθυντήριες γραμμές του 2006 να ενσωματώσουμε αυτό το πολύ ισχυρό μήνυμα, ότι δηλαδή όλα αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Και καλώς, αλλά ε, μένει η απόσταση να καλυφθεί. Για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο προτείνουμε να θέσουμε περιβαλλοντικούς στόχους και στόχους που έχουν να κάνουν με την αλλαγή του κλίματος, ε, στο πλαίσιο της ε, πρωτοβουλίας για συνολικά παγκόσμια δημόσια αγαθά. Θέλουμε δηλαδή το 25% των, ε, των κονδυλίων να ε, αφιερώνονται σε ε, προγράμματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον και την αλλαγή του κλίματος. Και βεβαίως υπάρχει και ο γενικότερος στόχος του 20% ως προς τις κλιματολογικές αλλαγές. Και όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται στα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα γεωγραφικά λοιπόν χρηματοδοτικά εργαλεία ε, θα συμπεριλάβουμε αυτό αυτό το ποσοστό του 25% και 20% αντιστοίχως. Ε, θα ε, ολοκληρώσω κάπου εδώ την παρουσίασή μου και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω ε, στις ερωτήσεις που τυχόν θα τεθούν. Ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στην κυρία Κέμφ για να απαντήσετε στα διάφορα ερωτήματα που σας έχουν θέσει. Ευχαριστώ όλους για τις ερωτήσεις σας. Δείχνετε ότι υπάρχει και γνώση και ενδιαφέρον για τη σχέση ανάμεσα στην ανάπτυξη και το περιβάλλον. Θα ξεκινήσω ανάποδα με την τελευταία ερώτηση για τη σχέση ανάμεσα στο μακροπρόθεσμο και στη μακροπρόθεσμη αηφορία και στα βράχη πρόθεσμα κέρδη θα έλεγα στην ανάπτυξη. Νομίζω ότι δώσατε πάνω κάτω οι ίδιοι την απάντηση λέγοντας ότι τίθεται εδώ ένα θέμα αντιτιθέμενων συμφερόντων. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε μέσω της Poverty Environmental Initiative είναι δύο πράγματα. Πρώτον, να ανεβάσουμε τα επίπεδα δυνατής προστασίας. Γιατί αν αναφερθούμε στα δικαιώματα στη υγεία, στα δικαιώματα στην καθαριότητα κτλ. θα δει κανεί ότι είναι μεσοπρόθεσμα μέσα τα οποία αφορούν τους φτωχούς πληθυσμούς κυρίως γιατί αυτοί είναι οι πληθυσμοί οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε νερό και σε υπηρεσίες υγείας ή μάλλον σε συνθήκες υγιεινής καλύτερα. Εάν οι φτωχοί λοιπόν δεν παίρνουν μέρος στη διαδικασία α, λήψεως αποφάσεων γιατί δεν συμμετέχουν εν πάση περιπτώσει στις διαδικασίες αυτές και δεν έχουν ταυτόχρονα και πρόσβαση σε πόρους όπως το θέμα της διαχείρισης των υδάτων, το θέμα της διαχείρισης των γεών, γιατί είναι φτωχοί και περιθωριοποιημένοι, είναι το πρώτο πρόβλημα, δηλαδή πώς θα πάρουν μέρος στη συζήτηση. Είναι ένα πρώτο βήμα. Πρέπει λοιπόν να τους εμπλέξουμε στις αξιολογήσεις και στις διαδικασίες ε, εφαρμογής των αποφάσεων, των ε, συνεπειών των αξιολογήσεων. Οπότε θα πρέπει να προσπαθήσουμε τα άμεσα οικονομικά κέρδη να μην επικρατήσουν εις βάρος της, της μακροπρόθεσμης αηφορίας. Εδώ οι εταίροι όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εσείς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορείτε να είσαστε ένα σημαντικός εταίρος για την μακροπρόθεσμη θα έλεγα ανάπτυξη και όχι για τις βραχυπρόθεσμες δράσεις. Τώρα για την πράσινη οικονομία. Είναι αυτό τρόπος να το πετύχει κανείς αυτό, αλλά δεν θα πρέπει να θεωρηθεί από τις φτωχές χώρες σαν εμπορικό εμπόδιο. Γιατί πολλές φτωχές χώρες θεωρούν ότι η συζήτηση για την πράσινη οικονομία είναι ένα επιπλέον εμπόδιο για την πρόσβασή τους στις αγορές. Και πιστεύουν ότι η ουσία της συζήτησης είναι το πώς μπορεί να έχει κανείς μια πράσινη οικονομία, μένει η οποία όμως να απασχολεί τον κόσμο ε, δεν μιλάμε εδώ για, κεφαλ, για εντατική χρήση κεφαλαίων, μιλάμε για εντατική χρήση ανθρώπινου δυναμικού. Το να βάζει κανείς πάρα πολλά λεφτά ας πούμε στην παραγωγή ε, ηλιακής ενέργειας είναι κάτι το οποίο οικολογικά είναι ενδιαφέρον, έχει όμως υψηλό κεφαλαιοκικό κόστος, δεν δημιουργεί θέσεις εργασίας, και οι τοπικοί κάτοικοι θα έλεγα δεν είναι σε θέση να πληρώσουν τις υπηρεσίες αυτές γιατί δεν έχουν τα απαιτούμενα εισοδήματα. Οπότε δεν έχουμε να κάνουμε με μια αηφόρο πηγή ενέργειας. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια πράσινη οικονομία η οποία να δίνει ευκαιρίες απασχόλησης στους κατοίκους μιας περιοχής, στους φτωχούς μιας περιοχής. Είναι το θέμα το οποίο μας απασχολεί. Ο κύριος αναφέρθηκε στο πώς μπορούμε να πείσουμε τις κυβερνήσεις των αναπτυσσομένων χωρών να περάσουν σε παραγωγές οι οποίες να είναι υπέρ των φτωχών, να δημιουργούν πολλές θέσεις απασχόλησης και να μην κόβουν και τα δάση τους. Πώς μπορούμε να πιέσουμε τις φτωχές αυτές χώρες να αναγνωρίσουν μακροπρόθεσμα τα ωφέλη για τους πληθυσμούς τους μέσω των μακροπρόθεσμων πολιτικών. Μία από τις λύσεις η οποία προτείνεται είναι το λεγόμενο σχέδιο πρόγραμμα UNEP-REP. Πληρώνουμε φτωχές κοινότητες να διατηρήσουν τα οικοσυστήματα. Σε αυτή τη φάση υπάρχουν κάποια τέτοια προγράμματα και στα Κονγκό και στο Βιετνάμ ε, η κοινότητα δεν ασχολείται με το να κόψει τα δέντρα, αλλά να διατηρήσει τις περιοχές οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν αργότερα για παραγωγή προσόδου προς τον τοπικό πληθυσμό, να χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα της δασοκονίας και έτσι θα προστατεύσουν και τη δική τους ευημερία. Και αυτό θα χρησιμοποιηθεί επίσης και για την αντιστάθμιση ε, ποσοτήτων εκπομπής διοξιδίου άνθρακα κτλ. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δούμε τα πράγματα από κάτω, από τη βάση, γιατί πρέπει να καλυφθούν οι ανάγκες της βάσης, ας πούμε, για καύσιμα από ξύλο και πρέπει να δώσουμε ε, οικονομικά μέσα στις κοινότητες ε, να σεβαστούν το περιβάλλον αλλά καλύπτοντας και τις ανάγκες τους και αυτό θα το καλύψουμε οικονομικά εμείς. Είναι λοιπόν μια καλή μέθοδος θα έλεγα αν μπορούν ε, να δούμε, να είμαστε σίγουροι ε, αν προτιμάμε να προωθήσουμε μια οικονομική δραστηριότητα όπου λίγοι κάτοικοι μιας περιοχής χρησιμοποιούν το δάσος για παραγωγή εσόδων ε, ή μακροπρόθεσμα να βοηθήσουμε τη διατήρηση του δάσους και την επιβίωση των πληθυσμών. Τώρα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τι μπορούμε να κάνουμε στην περίπτωση της Ρουάντας σαν παράδειγμα έτσι ώστε να παράγονται ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσω αναδασώσεων, μέσω καλής χρήσης των υδροτόπων κτλ. Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι έχουμε να κάνουμε με μια χώρα με μεγάλη πυκνότητα πληθυσμού. Κάθε τετραγωνικό εκατοστό χρησιμοποιείται για γεωργικούς λόγους έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες ε, τρόφιμα του πληθυσμού. Δεν υπάρχει λοιπόν πάρα πολλής χώρος για να φυτευτούν παραγωγές ανανεώσιμης ενέργειας που να οδηγούν στην ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το θέμα είναι να χρησιμοποιήσουν τα δάση τα οποία υπάρχουν και τα εδάφη τα οποία υπάρχουν με καλύτερο τρόπο. Να παράγουν περισσότερη υδροελοκτική ενέργεια, ε, να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές επιλογές. Πολλές από τις χώρες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα όταν περνούν σε ανανεώσιμες πηγές να βλέπουν τα κόστος των τροφίμων να αυξάνονται διότι περιορίζεται η αρρώσιμη γη για την παραγωγή των τροφίμων μέσω της καλλιέργειας ενεργειακών ε, φυτών. Πρέπει να δούμε λοιπόν ότι το σύστημα αυτό δεν είναι πάντα αηφόρο, τουλάχιστον σε επίπεδο χρήσης, όταν οι πόροι είναι περιορισμένοι. Και επειδή η Ρουάντα είναι μια μικρή χώρα, με, υψηλές, ε, με υψηλά ποσοστά καλλιεργούμενης γης. Η απόφαση αφορά την σωστή χρήση των ε, δασών και των υγροτόπων. Να περάσω τώρα σε μία ερώτηση του Ντίας Δεμέρα για το πώς λαμβάνουμε υπόψη μας κοινωνικές και εθνοτικές διαιρέσεις στα πλαίσια της αηφορίας ε, στο περιβάλλον. Πράγματι, ιστορικά ένα τμήμα του πληθυσμού είχε αποκλειστεί από τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες γιατί ήταν από τη μία πλευρά του εθνοτικού ρήγματος θα έλεγα. Στη Ρουάντα χρησιμοποιήθηκαν όμως οι αναπτυξιακές προσπάθειες για να ξεπεραστούν οι διαιρέσεις οι εθνοτικές. Η κυβέρνηση αυτή λέγει ότι τώρα είμαστε όλοι κάτοικοι της Ρουάντα, δεν υπάρχουν εθνικές καταβολές, τώρα στην πραγματικότητα τι συμβαίνει είναι άλλο θέμα. Αλλά όλοι μπορούν να είναι υπερήφανοι για την αναπτυξιακή ατζέντα και κάθε πολίτης μπορεί να ωφεληθεί από την ταχεία ανάπτυξη της ε, Ρουάντα και σε αυτή την περίπτωση οι εθνικέ οι εθνοτικές διαιρέσεις γίνονται λιγότερο σημαντικές. Αυτό υποτίθεται ότι προσπαθούν να κάνουν. τα αποτελέσματα σε επίπεδο ανάπτυξης είναι εντυπωσιακά. Αν πάτε αυτή τη στιγμή στην Ρουάντα, θα δείτε ότι οι καταστροφές που είχαν συμβεί το 2004 έχουν αρχίσει και καλύπτονται. Αυτό έχει οικονομικά ωφέλη, έχει όμως και πολιτικά προβλήματα, δημιουργούνται Υπάρχουν πάντα φυσικά τα υπέρ και τα κατά των αναπτυξιακών διαδικασιών, αλλά εάν πράγματι η ανάπτυξη βοηθήσει όλο τον κόσμο και τους φτωχούς, είναι σαφές ότι οι εθνοτικές διαιρέσεις μπορεί να βοηθηθεί να ξεπεραστούν. Και μετά μια άλλη ερώτηση για το εάν η ανάπτυξη καταστρέφει το περιβάλλον σε κάποιες χώρες οι οποίες μας έχουν δώσει το κακό παράδειγμα, Κίνα, Ινδία κτλ. Νομίζω ότι και εδώ μπορεί να περάσει κανείς από τα κάτω προς τα πάνω. Βασική ιδέα της πράσινης οικονομίας είναι να μπορέσει να χρησιμοποιήσει τις πολιτικές του για το περιβάλλον για να βγάλει τον κόσμο από τη φτώχεια. Το πώς λοιπόν μπορεί κανείς να περάσει ε, σε μια αναπτυξιακή πορεία είναι κάτι το οποίο πρέπει να αναζητήσουμε. Σαν παράδειγμα συνεργαζόμαστε ε, στο Μοντεβίντεο στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος με φτωχούς συλλέκτες σκουπιδιών, απορριμμάτων και τους, ε, ε, ρακοσυλλέκτες λοιπόν του Μοντεβιδέου τους βοηθάμε, βοηθάμε την κυβέρνηση να τους βοηθήσει και οι εκτιμήσεις τις οποίες κάνουμε τώρα είναι ότι μια κοινωνική ομάδα που προέρχεται από ένα πολύ χαμηλό θα έλεγα κοινωνικό στρώμα τώρα νιώθουν ένα κάποιο πνεύμα επιχειρηματικότητας γιατί πράγματι παρέχουν χρήσιμες υπηρεσίες και οικονομικά ωφέλιμες για αυτούς μέσω της ανακύκλωσης. Ε, ενισχύουν τη θέση τους, βοηθούν το περιβάλλον ε, δεν υπάρχουν εδώ ασυμβατότητες και νομίζω ότι από τα παραδείγματα αυτά μπορούμε να μάθουμε για να βοηθήσουμε τα πράγματα να πάνε καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν για αυτήν την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη παρουσίαση. Νομίζω ότι τις δημοσιεύσεις θα τις βρούμε φυσικά στις ιστοσελίδες σας. Θα περάσω τώρα στην Κάμπι Τσίμα, η οποία θα παρουσιάσει ε, κάποιες ε, περιπτώσεις ε, μελέτης του δεύτερου πάνελ. Thank you very much, Ska. Uh, first of all, Ευχαριστώ πολύ, Σκά. Θα ήθελα και εγώ από πλευρά μου να ευχαριστήσω για την παρουσίαση αλλά και για την διασύνδεση που παρουσιάσατε των συνεπειών της εκβιομηχάνησης με την καταστροφή των οικοσυστημάτων και της φτώχειας. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο εμείς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επικεντρωνόμαστε περισσότερο σε, αυτό το, σε αυτή τη σύνδεση αλλά και να αναλογιζόμαστε τι του στρατηγική εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσαμε φέρει πέρι στην αργιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαμε να σχεδιάσουμε κάτι διαφορετικά γιατί και τα αισθήματα που επισημάνατε εσείς προς τη χρήση των γεών, την κατάχρηση των ε, πόρων για την παραγωγή ε, ενέργειας είναι επισημάνσεις οι οποίες και την ε, πτυτικότητα των ε, τιμών των τροφίμων μπορούν να επηρεάσουν. Και τώρα, τώρα θα ήθελα να καλωσορίσω και τους νεαρούς επισκέπτες μας εδώ που κάθονται στο πίσω μέρος της αίθουσας και να περάσουμε στο θέμα των ε, πρακτικών μελετών που δείχνουν ε, περιβαλλοντικές σχέσεις και δραστηριότητες. Δυστυχώ δεν μπορούσαμε να έχουμε ένα ηχητικό υλικό που θα μπορούσε να παρουσιάσει μια μελέτη για την, ε, τις συνέπειες των τοξικών υλών που θα ήταν πολύ χρήσιμο να ακούσουμε. Θα κοιτάξουμε να δούμε αν μπορούμε να την φέρουμε κάποια άλλη στιγμή στην επικαιρότητα. Παρακαλώ τώρα τον κύριο Williams, επικεφαλής ε, του τμήματος φίλη της γης Νιγερία. που έχει και ως ε, δικηγόρος δραστηριοποιηθεί στις ε, περιβαλλοντικές ε, αγωγές, μαζικές αγωγές έχει ιδιαίτερα αγωνιστεί για την αλλαγή στη Δυτική Αφρική και ειδικότερα την Ιγυρία της, ε, του τρόπου διαχείρισης των ε, απορριμμάτων και κυρίως ε, και γενικότερα την προσέγγιση του περιβάλλοντος. Το θέμα του λοιπόν είναι η συνέπειες των δραστηριοτήτων των πετρελαϊκών εταιριών ως προς το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την ανάπτυξη στην υποσαχάρη Αφρική, το δέλτα του Νίγηρα. Κύριε Πρίνς Τσίμα Βίλιαμς, παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ξιότιμες κυρίες και κύριοι, βουλευτές, συνάδελφοι. Κυρίες και κύριοι, μεγάλη η τιμή που μου κάνετε να με υποδέχεστε μεταξύ σας για να συζητήσω ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις δραστηριότητες των πετρελαϊκών επιχειρήσεων, εταιριών και τις συνέπειες αυτών στο περιβάλλον στην, στο Δέλτα του Νείλου. Έχω μια παρουσίαση, μάλλον όμως ο χρόνος δεν μου αρκεί για να την ε, παρουσιάσω διεξοδικά. Θα προτιμούσα να συζητήσουμε τα θέματα, θα ήταν πολύ πιο ενδιαφέρον φαντάζομαι για όλους. Και δεν ήθελα ξεκινώντας να πω ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της καταστροφής του οικοσυστήματος του Δέλτα του Νείλου προκύπτει από τις δραστηριότητες πετρελαϊκών εταιριών, εταιριών φυσικού αερίου ε, στην περιοχή μας, προερχομένων όμως από την Ευρώπη και κυρίως οι μεγάλες εταιρείε όπως η Shell, η Agip, NI Agip, και βέβαια αντίστοιχα αμερικανικής πρόλευσης εταιρείε και λοιπές. Όπως σας είπα, δεν θα εκφωνήσω την ομιλία που είχα υπόψη. Θέλω μια γενική συζήτηση να κάνουμε για τις δραστηριότητες των πετρελαϊκών εταιριών και τη φτώχεια. Ας κοιτάξουμε λοιπόν τις συνέπειες στο Δέλτα του Νείλου των δραστηριότητων αυτών. κατάσταση είναι μάλλον δύσκολη για τους πολίτες που ζουν στο Δέλτα του Νίλου του Νίγηρα. Διότι ενώ θα έπρεπε να είναι ευλογία τα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, τελικά μετατρέπονται σε πληγή σε ζημιά για το λαό μας. Οι πολίτες της Νιγερίας και όσοι ζουν στο Δέλτο του Νίγηρα ιδιαίτερα Βεβαίως αναγνωρίζουν ότι ε, κερδίζουν πολλά, κερδίζει πολλά, ιδιαίτερα η, η οικονομία του κράτους της Νιγηρίας από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, αλλά ο κοινός πολίτης στην καθημερινή του ζωή, αυτό που γνωρίζει, πάνω απ' όλα είναι η μόλυνση, η ρήπανση που φέρνει η εξόριξη του πετρελαίου και του φυσικού αέριου. Θα μπορούσα να σας δώσω μια περιγραφή Θα μπορούσα να δώσω πολλά παραδείγματα ε, της καταστροφής που φέρνει το πετρέλαιο, η εξόρυξη του πετρελαίου από μόλυνση, ρήπανση, ζημιές, προβλήματα τα οποία προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε στο Δέλτα του Νίγηρα. Ακόμη και πετρελαιοκυλίδες που έχουν καταστρέψει ευρείς περιοχές του Δέλτα του Νίγηρα. Αλλά θα σας πω μόνο το εξής. Ανάμεσα στο Δεκέμβριο πέρσι και τον Ιανουάριο εφέτος είχαμε καταστροφικές καταστροφικά ε, ατυχήματα τα οποία είχαν παγκόσμια εμβέλεια και τεράστιες επιπτώσεις στην περιοχή του Δέλτα του Νίγηρα. Ιδιαίτερα στις 26 Δεκεμβρίου του 2011 η πετρελοκυλίδα από την περιοχή Μπούγκα της ε, Σέλα, της ε, του, της περιοχής εξόρυξης ε, της Shell μέσα στη θάλασσα. Μια εξέδρα η οποία αξιοποιείται ιδιαίτερα, το προϊόν της δηλαδή αξιοποιείται ιδιαίτερα για εξαγωγές προς την Ευρώπη, είχε κατά τη μεταφορά από την πλατφόρμα ε, σε δεξαμενόπλιο επί της θαλάσσης ε, του πετρελαίου υπήρξε διαρροή με μια πετρελοκυλίδα λίδα η οποία επηρέασε τη ζωή των παράκτιων κοινοτήτων και συνολικά εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών. Πριν έρθω εδώ, την Ένωση των Αριστεχνών Αλλιέων της ε, Νιγηρίας. από περιοχές παράκτιες και παρόχθιες, οι οποίοι ήρθαν και μου ζήτησαν να τους βοηθήσω στον αγώνα τους κατά της ΣΕΛ και κατά της πετρελοκυλίδας Μπούγκα. Είναι πάνω από 20.000 αυτοί οι οποίοι έχουν χάσει την πηγή εισοδήματος τους που αντλούσαν από τη θάλασσα λόγω αυτής της πετρελαιοκυλίδας. Διότι λόγω της τάσης της ΣΕΛ και των ε, Νιγηριανών αρχών δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν καν τα ύδατα της περιοχής. Από το Δεκέμβριο λοιπόν μέχρι τώρα, καθώς δεν έχει καθαριστεί αυτή η πετρελαιοκυλίδα, δεν έχουν εισοδήματα, δεν έχουν καμία πηγή εσόδων και δεν έχουν καν δουλειά, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει κάτι τέτοιο. Τι κατάσταση μπορεί να προκαλέσει και το να μείνει κανεί σε υποχρεωτική ε, ανεργία γιατί δεν έχει αντικείμενο εργασία, αλλά έχει, ε, ταυτόχρονα έχει χάσει και το εισόδημά του, δεν μπορεί να ταΐσει την οικογένειά του και δεν ξέρει πού μπορεί να στραφεί. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πολύ μεγάλη αποσταθεροποίηση, αστάθεια και βέβαια αποτελεί και το επίκεντρο των προβλημάτων που γνωρίζουμε στο Δέλτα του Νίγηρα. Και αυτό βέβαια μπορεί να οδηγήσει σε πολύ σημαντικές, πολύ, πολύ ε, σοβαρά ψυχολογικά ε, ζητήματα και προβλήματα υγείας. Αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα. Η πετρελοπληγίδα Μπούγκα. Και χαίρομαι που είναι εδώ η κυρία Κέμφ, διότι το πρόγραμμα για το περιβάλλον των Ηνωμένων έχει εκδώσει μια ε, έκθεση η οποία εμάς, εμένα ως ε, αγωνιστή για το περιβάλλον, ως ακτιβιστή, δεν με εξέπληξε πρέπει να πω, γνωρίζοντα τα πράγματα στην ε, περιοχή αυτή. Γνωρίζουμε λοιπόν όλοι και πρέπει να γνωρίζουν και οι βουλευτές φαντάζομαι ότι πριν την έρευνα του περιβάλλοντος αυτής της της, ε, του προγράμματος περιβάλλοντος, εμείς αντιταχθήκαμε στο επιχείρημα ότι η Shell έχει καταστρέψει την Ουγκούνιλάντ, ε, την Ουκουλιλάνδη και θα έπρεπε να επανέλθει σε αυτήν και όπου η κυβέρνηση θα προσπαθούσε να βοηθήσει να επανέλθει η Shell. Δεν έχει κανείς δηλαδή ε, το δικαίωμα δεοντολογικά να προσβάλλει, να αμφισβητήσει μάλλον τα Ηνωμένα Έθνη και ως εκ τούτου εάν τα Ηνωμένα Έθνη πούν ότι μπορεί να επανέλθει η Shell στην περιοχή αυτή, αν δηλαδή το πρόγραμμα για το περιβάλλον μπορούν να πούν ότι είναι εντάξει, τότε και ο λαός σεβόμενος τα Ηνωμένα Έθνη θα αποδεχθεί την πρόταση αυτή. Η έκθεση υπευλάθη στον ε, πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Νιγηρίας πριν από 8 μήνες με συστάσεις. Μια έκθεση η οποία λέει ότι η Γκουνιλάνδη έχει τόσο πολύ ρήπανση υποστεί που θα χρειαστούν ακόμα και 30 χρόνια για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Ακόμη και άμεση δράση αποκατάστασης που είχε συσταθεί από την έκθεση πριν από έξι μήνε, όπω είπα, και περισσότερο από έξι μήνε που είχε υποβληθεί η έκθεση. Έχουν περάσει 6 μήνε λοιπόν, 8 μήνε και δεν έχει γίνει τίποτα. Ένα πολύ ωραίο έγγραφο ήταν αυτή η έκθεση. Τουλάχιστον εμά ε, μα προσέφερε όπλα κατά τη κυβέρνηση για να επιβεβαιώσουμε ότι αυτό το οποίο λέμε και διεκδικούμε είναι σωστό. Αλλά τι να την κάνουμε μια έκθεση. Άλλο ένα μπόδι μπροστά μας, άλλη μια πρόκληση μπροστά μας για δε την κυβέρνηση η δουλειά είναι πάντα ίδια, δεν αλλάζουν τίποτα. Θέσπισαν τελευταία περίοδο τρεις ε, επιτροπές σε ομοσπονδιακό επίπεδο με στόχο την μελέτη της έκθεσης ε, του προγράμματος για το περιβάλλον των Ηνωμένων Εθνών που και πάλι καταλήγουν στην, ε, στα συρτάρια του Υπουργού Πετρελαίου που είναι πρώην διευθυντής της ΣΕΛ στην Ιγυρία. Καταλαβαίνετε βέβαια τι είδους τύχη θα έχει μια τέτοια εταιρεία. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή τη μοίρα είχε η έκθεση της ΣΟΝΕΠ ε, για την Ουγουνιλάνδη. Αντίστοιχα και σε άλλες περιπτώσεις βέβαια στο Δέλτα του Νίγηρα γιατί δεν ήταν ε, μόνο η Ουγουνιλάνδη εκείνη η οποία υπέστη πετρελοκύλη. Δεν είναι πολλά άλλα σημεία της, ε, του Δέλτα του Νίγηρα. Το 1998 ε, μία από τις μεγαλύτερες πετρελοκυλίδες από την Exxon Mobil και την πλατφόρμα Ιντόχο. ...24.000 ε, ε, βαρέλια κατέργασης του πετρελαίου έφτασαν στη θάλασσα. Αντίστοιχη καταστροφή με αυτή της πετρελοκυλίδας Μπούγκα. 40.000 βαρέλια λένε, αλλά είναι πολύ μεγαλύτερη πετρελοκυλίδα από αυτό και δεν υπάρχει τρόπος επαλήθευση της πραγματικής ποσότητας του πετρελαίου που ε, χύθηκε στη θάλασσα και των συνεπειών αυτού. Τουλάχιστον λοιπόν η πετρελοκυλίδα Μπούγκα καταγράφηκε ω προ τι συνέπειε τη μέσα μια έκθεση του προγράμματο για το περιβάλλον των Εθνών. Είχαμε όμω στι αρχέ του χρόνου και άλλη κοιλίδα από την Σευρών αυτή τη φορά. Μια έκρηξη σε μια μονάδα εξόρισης, πάλι πλατφόρμα στην ανοιχτή θάλασσα, όπου εμείς είχαμε αγωνιστεί βέβαια και ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίου είχαμε σταθεί κατά της έκθεσης ε, τη ΣΟΝΕΠ γιατί λέγαμε ότι είναι ξεκάθαροι λόγοι. Η αγωγή, η πετρελαιοαγωγή που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις, οι εταιρείε αυτές είναι πολύ παλιοί. Πολλοί έχουν εξαντλήσει πλέον και το, ε, τη διάρκεια ζωή του. Και έτσι με την ελάχιστη επιπλέον πίεση ε, σκάνε. Και ζητήσαμε μια επαλήθευση της αντοχής αυτών των ε, εγκαταστάσεων μεταφοράς του πετρελαίου που όμως δεν πραγματοποιήθηκε και έτσι στην περίπτωση της Ευρών ε, έσκασε ο αγωγός μας είπαν ότι έφταιγε η υψηλή πίεση ε, κατά την ροή του πετρελαίου σε ένα παλαιό αγωγό. Από τα μέσα Ιανουαρίου που ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά δεν έχει σταματήσει ακόμα. 10 χιλιόμετρα στα ανοιχτά των ακτών. Μένεται μια πυρκαγιά εδώ και εβδομάδες, δεν μπορεί κανείς να κάνει τίποτα και ο λαός δεν έχει να ζήσει πια, δεν μπορείτε το νερό να πιει. Εξαρτάται όλος ο πληθυσμός της περιοχής ακόμα και για τις ε, πηγές πόσιμου νερού από, την, ε, από τον ε, ορίζοντα της περιοχής. Κάποιοι το πίνουν το νερό μια και δεν έχουν καμία άλλη λύση. Κάποιοι που πείθουμε ότι είναι μολυσμένο το νερό. Βέβαια η Σευρών αρχικά υπεστήριξε ότι δεν υπήρξε καμία ε, ζημιά στο περιβάλλον. Αλλά βέβαια η οργάνωσή μου με μελέτη που έκανε πιτόπου στην περιοχή απέδειξε όχι μόνο τη σημαντική ρήπανση αλλά και τις σημαντικές καταστροφές στην, ε, ε, στα θαλάσσια είδη, στα, στο ζωικό βασίλειο της περιοχής που βεβαιώσε και μια αντίστοιχη έρευνα και ντοκιμαντέρ του BBC. Αυτή είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της Νιγηρίας που ζουν στο Δέλτα του Νίγηρα ο Νομπίτο Μπάση που είναι ορμόδιο για τα θέματα αυτά Μα λέει ότι στην έκθεση UNEP κάποιε προτάσει θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι ο κόσμο στην ε, περιοχή μα γεννιέται μέσα στη μόλυνση, ζει όλη του τη ζωή μέσα στη μόλυνση, πεθαίνει μέσα στη μόλυνση και δεν έχει καμιά διέξοδο από τη ρήπανση αυτή διότι είναι τόσο κατεστραμμένο το οικοσύστημα στην περιοχή του. Αυτά μόνο οι πετρολοκυλίδες. Ε, αντίστοιχα το φυσικό αέριο και μέθοδοι ε, που ε, χρησιμοποιούνται στην περιοχή μας αλλά απαγορεύεται να υπάρχουν στην Ευρώπη, Δυτική Ευρώπη είναι παράνομες, ωστόσο στην Ιγυρία συνεχίζονται το λεγόμενο flaring του αερίου, φυσικού αερίου, το οποίο ε, προξενεί τεράστια ζημιά στο περιβάλλον. Και όμω είναι ανεκτό από την κυβέρνηση, διότι αυτή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό για τα έσοδά τη από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Ε, Εμεί όμω δεν ε, θεωρούμε ότι πρέπει αυτό να αποτελεί λόγο να παραβλέψουμε την ε, σοβαρή ζημιά στο περιβάλλον που μπορεί να προκαλέσει αυτή η μέθοδος του flaring. Γιατί θα πρέπει να βρεθεί μια άλλη λύση και ε, με την ε, πιθανολόγηση απαγόρευσης του φλέρινγκ αυτού μπορούμε να αναστήσουμε διαφορετικές λύσεις. Η Ιγυρία είναι από τις χώρες οι οποίες έχει τους μεγαλύτερους πόρους ε, ε, σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, αλλά λόγω της ανάφλεξης αυτής ε, του flaring χάνει πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο. από τις ειδήσει να παρακολουθήσατε ε, Τι μεγάλες διαδηλώσει και τα συλλαλητήρια που έγιναν στους δρόμους της Νιγηρίας λόγω τη επιδότησης που προσφέρει η κυβέρνηση για το φλερινγκ 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια επιτρέπει η κυβέρνηση να χάνονται κάθε χρόνο λόγω αυτής της ανάφλεξη του φυσικού αερίου με αποτέλεσμα να πληρώνουμε όλοι πιο ακριβή τιμή. Και βεβαίω δημιουργείται μια κατάσταση κρίσης. Είτε υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνη μεταξύ πολιτών και κυβέρνησης και των μεγάλων ε, πολιεθνικών από την άλλη, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, είναι σαφές ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις δηλώνουν εκατομμύρια δολάρια ε, κέρδη από το πετρέλαιο. Από πού όμως προέρχονται και τι παίρνουν για αντάλλαγμα καταστρέφεται το περιβάλλον, καταστρέφεται ο κοινωνικός ιστός, δημιουργούνται προβλήματα με όλα αυτά τα επεισόδια ανάφλεξης αερίου. Η ανάφλεξη αερίου προκαλεί τεράστια προβλήματα στην υγεία και βεβαίως ε, επιτείνει την αλλαγή του κλίματος και όλα αυτά έχουν ε, επιβεβαιωθεί επιστημονικά. Στην Ιγυρία Έχουν υπάρξει δικαστικές αποφάσεις που καταδικάζουν την ανάφλεξη του αερίου, την καθιστούν παράνομη και διατάζουν ε, την Shell και τις άλλες εταιρείες να σταματήσουν αυτή την πρακτική άμεσα. Παρ' όλα αυτά το συνεχίζουν οι εταιρείες αυτό. Οφείλουν οι εταιρείες να δώσουν προθεσμίες και συνεχίζουν να δίνουν προθεσμίες στην κυβέρνηση κατά πώς νομίζουν. Και η κυβέρνηση συνεχίζει να συνεργάζεται με αυτές. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά αβέβαιη, Γιατί υποτίθεται ότι, τα... ότι η κυβέρνηση υποτίθεται ότι πρέπει να υπερασπίζει τα συμφέροντα των πολιτών. Ωστόσο, το 2010 η κυβέρνηση προσπαθούσε να ψηφίσει σχετικό νόμο για το πετρέλαιο στην Ιγυρία, ρυθμίζοντας όλες τις δραστηριότητες. Σε αυτό το πλαίσιο ε, έγινε επαναδιαπραγμάτευση και επανασχεδιασμός των ε, συμπράξεων, έτσι ώστε τελικά οι μεγάλες εταιρείες έδρασαν κατά τρόπο ώστε το τελικό νομοσχέδιο να είναι διατυπωμένο κατά πώς του συμφέρει ή να μην ψηφιστεί, να μην περάσει καθόλου. Δεν έχει λοιπόν εγκριθεί το σχετικό νομοσχέδιο. Γίνεται ακόμα διαπραγμάτευση Και βεβαίως η διαπραγμάτευση γίνεται μέσα σε μια επιτροπή στην οποία ε, συμμετέχει και ο Υπουργό ε, περί πετρελαϊκών θεμάτων τη κυβέρνηση, ο οποίο είναι και πρώην διευθυντή τη ΣΕΛ ούτω ή άλλω. Βλέπετε τα προβλήματα λοιπόν. Ας περάσουμε τώρα στις συνέπειες. Ποιε είναι οι συνέπειες. Στο Δέλτα του Νίγηρα έχουμε, είμαστε μάρτυρες ε, στρατιωτικών δράσεων θα έλεγα, εκρήξεις, απαγωγές είναι πράγματα που συμβαίνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ως περιβαλλοντολόγος εγώ καταδικάζω τέτοιου είδους δράσεις. Καταδικάζω απερίφραστα όλες αυτές τις ε, δράσεις και το έχω επαναλάβει και εντός Νιγηρίας και εκτός. Σε όλα τα φόρουμ που έχω παραστεί, τέτοιου είδους καταστροφές των εγκαταστάσεων των εταιριών δεν πρόκειται να ε, λύσουν τα προβλήματά μας. Οι εγκληματικές δραστηριότητες δεν πρόκειται να λύσουν τα προβλήματά μας, αντιθέτως θα μας δημιουργήσουν ακόμα περισσότερα. Αυτό το έχω επαναλάβει εγώ πολλές φορές. Θα πρέπει να έχουμε άμεσους συνομιλητές και να δημιουργηθεί μια κατάσταση κατά την οποία όλοι θα σέβονται τα δικαιώματα και θα εφαρμόζουν τις αξίες που ε, ενστερνιζόμαστε όλοι. Και γι' αυτό το λόγο άλλωστε η παρουσία μου εδώ σε αυτή την ακρόαση ε, είναι εξαιρετικά σημαντική για μένα τουλάχιστον διότι δεν θέλω να μιλώ μόνο για τα προβλήματα θέλω να αναφέρομαι και στις λύσεις. Ε, σε ποιες λύσεις μπορούμε να καταλήξουμε όλοι μαζί. Ποιες είναι οι λύσεις που συλλογικά μπορούμε να προσφέρουμε. Τα αιτήματα λοιπόν που υποβάλλω εδώ ε, είναι ουσιαστικά εκκλήσεις που έχω επαναλάβει ε, και στο παρελθόν σε διάφορα φόρουμ και στον ε, Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και σε, διάφορα άλλα, σε διάφορες άλλες ευκαιρίες σε διεθνείς διασκέψεις. Παρακαλώ λοιπόν να βοηθήσετε την Ιγυρία. Η Ιγυρία είναι αβοήθητη αυτή τη στιγμή. Χρειαζόμαστε βοήθεια. Εμείς ως Νιγηριανοί δεν μπορούμε να σταματήσουμε τους μεγιστάνες του πετρελαίου ούτως ώστε να μην καταστρέφουν το περιβάλλον μας, να μην δημιουργούν καταστάσεις κρίσης και να μην υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής μας. Βεβαίως έχουν γίνει ε, εκστρατείες κατά της περιβαλλοντικής ε, καταστροφής της Ογονιλάνδης ε, και γνωρίζουμε τελικά ε, ε, ποιοι ήταν οι υπέρμαχοι αυτών των εκστρατιών και ποια ήταν η κατάληξή τους. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν έχω να υποβάλω το εξή αίτημα. Καταρχάς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να βοηθήσει την Ιγυρία. Εξαναγκάζοντας τα κράτη-μέλη να ε, πείσουν και να επιβάλλουν στις εταιρείες τους να εφαρμόζουν τα ίδια πρότυπα παντού όπου έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα. Τα πρότυπα δηλαδή που ισχύουν και ε, στην χώρα προέλευσής τους. Να τα εφαρμόζουν και στη χώρα υποδοχής και να δοθεί βεβαίως χρηματοδοτική βοήθεια υποστήριξη κάθε είδους στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. ούτως ώστε να υπάρξει περισσότερη καταπολέμηση της καταστρατήγησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα μέσα και τα όργανα που έχει, ε, ε, ούτως ώστε να στηρίξει ε, την δημιουργία περιβαλλοντικών δικαστηρίων από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, όπου θα δικαστούν τα αδικήματα που έχουν διαπραχθεί καταστροφής του περιβάλλοντος, τα οποία και μπορούν να χαρακτηριστούν ως περιβαλλοντική γενοκτονία. Και αυτό το αίτημα το έχω υποβάλει και στον ε, διεθνή, ε, στην, και τον ε, Διεθνή Δικηγορικό Σύλλογο, στο Διεθνές Συνέδριο που είχε οργανώσει ο Διεθνής Δικηγορικός ε, Σύλλογος το 2011, Ούτω ώστε τελικά να τύχει στήριξη η έκκληση αυτή ε, στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Πιστεύω ότι αν το δεχθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό, θα αποκτήσει μεγάλη ισχύ αυτό το κίνημα στους κόλπους του ΟΗΕ για την σύσταση περιβαλλοντικών δικαστηρίων δηλαδή. Τρίτη έκκληση που απευθύνω. είναι η εξής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να υιοθετήσει κανονισμούς έτσι ώστε να είναι υποχρεωτικό οι εταιρείε ε, που δραστηριοποιούνται να πρέπει να απαντούν και να υπερασπίζονται τον εαυτό τους ενώπιον δικαστηρίων στις χώρες υποδοχής. Το Ολλανδικό Κοινοβούλιο είχε εξετάσει μια παρεμφερή ρύθμιση και θα, προσπαθήσω, ε, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε συνέχεια σε αυτή την προσπάθεια. Και τέλος, Θέλω να σας μιλήσω για κάτι που ε, ανέφερε και η κυρία Κέμφ και το, το παρατήρησα με μεγάλη χαρά. Ε, δηλαδή ε, για το γεγονός ότι οι κοινότητες ζουν από τα δάση τους και πρέπει να υποστηρίζονται σε αυτή την προσπάθεια. Όταν αν δούμε τη γενικότερη κατάσταση στην Ιγυρία, συμπεραίνουμε ότι τελικά καταλήξαμε στην τελευταία επιλογή. Είναι το Έτοιμά μας δηλαδή, αν αποτύχουν όλα ε, τα άλλα, να τύχουμε στήριξη. Εάν υπάρχουν νέα κοιτάσματα και βρεθούν νέα πετρελαϊκά κοιτάσματα. Ζητούμε να παραμείνουν εκεί στο έδαφος. Αν αφήσουμε το πετρέλαιο στο έδαφος, δεν θα υπάρχει πλέον καταστροφή. μπορούμε να έχουμε ένα ε, πρόγραμμα, ένα μηχανισμό για την καθαρή ανάπτυξη και βάσει του πρωτοκόλλου του Κιώτου να ανταλλάσσονται επιστώσεις αναφορικά με το ενεργειακό αποτύπωμα. Ε, θα σταματήσω κάπου εδώ και είμαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, λέει Πρόεδρος. Ευχαριστούμε τον κύριο Williams για αυτή την πολύ εντυπωσιακή παρουσίαση, πολύ λεπτομερή πολύ συγκεκριμένη. Σίγουρα εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούμε να διαδραματίσουμε έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Μπορούμε να συγκεντρώσουμε ε, τις πληροφορίες που μας δίνεται και να τις ε, ε, δημοσιοποιήσουμε, να τις δημοσιεύσουμε, ούτως ώστε ε, να γίνει μια δημόσια συζήτηση για τα προβλήματα της Νιγηρίας. Σίγουρα μπορούμε να κάνουμε περισσότερα και πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Και σίγουρα είναι σημαντικό να επαναλαμβάνουμε ότι οι επενδυτές ε, βεβαίως επηρεάζουν θετικά την ανάπτυξη στη χώρα στην οποία επενδύουν, ωστόσο μπορεί να έχουν και αρνητικές συνέπειες Είναι υπεύθυνοι λοιπόν οι επενδυτές αλλά και οι εθνικές ε, αρχές σε κάθε χώρα είναι πολύ υπεύθυνε ε, όταν επιλέγουν σε ποιον θα ε, δώσουν τη γη, θα την μισθώσουν ή θα την παραχωρήσουν για να αξιοποιηθούν τα εκάστοτε κοιτάσματα ή εκάστοτε πηγές. Οι ευθύνε λοιπόν των εθνικών αρχών είναι πολύ μεγάλες. Να δώσω τώρα το λόγο στους συναδέλφους. Παρακαλώ να είστε σύντομοι στις ερωτήσεις και στα σχόλιά σας προς τον κύριο Williams. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Βίλε και μετά τον κύριο Γκέρενς. Δεν θέλω να σας καθυστερήσω. Ο Βίλιος αναφέρθηκε στον Σκέν Σαροβίλα υπάρχει ένα θέμα. Σκοτώθηκε πριν κάποιες δεκαετίες. Ήμουνα τότε βουλευτής στην Κάτω Βουλή και 17 χρόνια μετά αναρωτιέμαι τι μπορούμε να πούμε. Δυστυχώς η κατάσταση είναι εξίσου κακή. Αυτό είναι απαράδεκτο. Ευχαριστώ κύριε Ντίβο, κύριε Γκέρντς. να ευχαριστήσω τον κύριο Williams για την παρουσίασή του, η οποία έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αναφέρεται σε ένα πραγματικό σκάνδαλο. Το σκάνδαλο έγκυται στο ότι οι, αρχές, ε, θα έλεγα η κυβέρνηση της Νιγηρίας ε, στην ουσία έχει παραμεριστεί από τις εταιρείες πριν εμπλακείς, εμπλακούν μάλλον σε κάποια εκμετάλλευση ε, πετρελαϊκού τύπου πρέπει να πάρουν μια αδειοδότηση. Αυτές οι αδειοδοτήσεις μπορεί να αφαιρεθούν, να ακυρωθούν αν οι συνθήκες οι οποίες ήταν προϋπόθεση δεν γίνονται αντικείμενο σεβασμού από την επιχείρηση. Έτσι πρέπει να είναι. Αν κάνω λάθος, αν δεν ανταποκρίνεται αυτό που λέω στην πραγματικότητα, διορθώστε με. Εφόσον ισχύει λοιπόν κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνει ό,τι δυνατόν έτσι ώστε η εξουσία του κράτους, η αρμοδιότητα η κρατική που έχει εκδώσει την άδεια πρέπει να γίνει σεβαστή. Ε, κατανοώ ιδιαίτερα αυτά που είπατε για ένα διεθνές δικαστήριο, τα σχετικά με ένα διεθνές δικαστήριο που θα μπορούσε να ασχοληθεί με τέτοιου είδους ε, καταστάσεις. Βέβαια διστάζω κιόλας λίγο διστάζω να το στηρίξω ήδη στα πλαίσια ενός ψηφίσματος γιατί αυτό θα μπορούσε να είναι και ένα νέο στάδιο το οποίο να αποδεικνύει και να επιβεβαιεί αν θέλετε την εξασθένηση της, των αρχών του κράτους ε, στο εσωτερικό του οποίου ε, εξελίσσεται αυτό το σκάνδαλο. Εμείς θέλουμε ισχυρές κυβερνήσεις αφρικανικές να γίνονται σεβαστές. Το κράτος δικαίου πρέπει να γίνεται σεβαστό, όπως είναι και προϋπόθεση στα πλαίσια της Συμφωνίας Κοτονού. Θα έλεγα επίσης ότι αντί να περάσουμε σε ψήφισμα, ίσως θα πρέπει να το συζητήσουμε, ζητώντας και την άποψη νομομαθών, εμπειρογνωμόνων μάλιστα στον τομέα του διεθνούς περιβαλλοντικού δικαίου και γιατί όχι να κάνουμε και μια έκθεση μια έκθεση η οποία θα έχει τη φιλοδοξία να, να επεξεργαστεί το θέμα το οποίο είναι πράγματι τεράστιο και όλα αυτά τα χρήματα τα οποία στην ουσία γίνονται αντικείμενο κατάχρησης, οι φυσικοί πόροι οι οποίοι αφαιρούνται από αυτούς οι οποίοι ηθικά και νομικά είναι κάτοχοι και τα έχουν, κάτοχοι και τα έχουν ανάγκη, και πρέπει να λυθεί ένα τέτοιο πρόβλημα γιατί αλλιώς στην ουσία εξασθενούμε τις αναπτυξιακές δυνατότητες των χωρών αυτών. Αλλά στην ουσία αυτό που ζητάμε σε μια πρώτη φάση είναι η αποκατάσταση των εθνική της εθνικής κυριαρχίας. Δεν ξέρω αν μπορείτε να σχολιάσετε αυτό το οποίο είπα και αν ανταποκρίνετε αυτό το οποίο είπα στην πραγματικότητα και σας καλύπτει κατά κάποιο τρόπο. Θα προτείνω να δώσω το λόγο και σε άλλους συναδέλφους να κάνουν τα σύντομα σχόλιά τους και στο τέλος να πάρετε το λόγο. Και έλα. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Συμμερίζομαι τις ανησυχίες σας για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος Βλέπουμε ότι και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εμπλέκονται σε τέτοιες διαδικασίες και είναι προβληματικό γιατί ακολουθούν και σέβονται κάποιους κανόνες περιβαλλοντικού στην Ένωση, αλλά όχι εκτός. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα σε όλο τον κόσμο και στη Λατινική Αμερική. Επιχειρήσεις έχουν την τεχνολογία να σεβαστούν τα υψηλότερα ή λιγότερο υψηλά περιβαλλοντικά κριτήρια, αλλά τα οποία τα ξεχνάνε όταν δραστηριοποιούνται σε άλλες περιοχές. Έχετε κάποιες πιο συγκεκριμένες προτάσεις για το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς σαν κοινοβούλιο. Αναφερθήκατε στη δυνατότητα δημιουργίας δικαστικών μέσων, αλλά έχετε κάποιες πιο συγκεκριμένες προτάσεις να μας κάνετε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κορτές Λάστρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Βίλιαμς που ήρθε εδώ στην ακρόαση αυτή. Είναι ένα θέμα για το οποίο έχουμε διαβάσει, είναι ένα θέμα το οποίο γνωρίζαμε. Ωστόσο, μας ε, έδωσε πολύ πρόσφατες πληροφορίες, νέα ενημερωτικά στοιχεία για το τι ε, συμβαίνει στο Δέλτα του Νίγηρα. Έχω δύο ερωτήματα να θέσω στον κύριο Williams, αλλά και στην εκπρόσωπο από το περιβαλλοντικό πρόγραμμα του ΟΗΕ. Καταρχάς, το θέμα της ε, κοινωνίας των πολιτών στο Δέλτα του Νίγηρα. το γεγονός ότι βιώνει αυτή τη δραματική κατάσταση. η οποία είναι πραγματικά ε, φοβερή και το έχουμε δει και με τα ατυχήματα που έχουν συμβεί στα πετρελαιοφόρα, στα δεξαμενόπλια ανά τον κόσμο. Πώς οργανώνεται η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, ποιες είναι οι πιέσεις που τους έχουν ασκηθεί, ε, πώς τις διαχειρίζεται, πώς ανθίσταται σε αυτές. Αυτό καταρχάς. Κατά δεύτερο λόγο, η τρίτη πρόταση που μας κάνατε, να πληρώνονται οι κοινότητες για να διατηρούν τα δάση και να μην τα κόβουν τα ε, δέντρα σε ορισμένες περιοχές. Θυμάμαι το Γιασούνι στον Ισημερινό είναι μία από τις περιοχές με τη μεγαλύτερη βιοπικιλότητα στον κόσμο και η κυβέρνηση του Ισημερινού μέσα από τον ΟΗΕ προτείνει την μη αξιοποίηση των πετρελαϊκών κοιτασμάτων σε αυτή την περιοχή προκειμένου να προστατευτούν οι φυσικοί πόροι και το περιβάλλον ε, με αντάλλαγμα μία οικονομική συγκεκριμένη αποζημίωση και του καθεξής. Θα μπορούσαμε λοιπόν επιλεκτικά ε, να διαλέξουμε κάποιες περιοχές ανά το κόσμο όπου να εφαρμόσουμε ένα τέτοιο σύστημα για λόγους εξαίρετου φυσικού κάλους να ε, θεωρήσουμε δηλαδή ότι δεν θα πρέπει να αξιοποιούνται τα κοιτάσματα ε, σε αυτές τις περιοχές και καλό θα ήταν να ε, χαράξουμε πολιτική, να εφαρμοστεί πολιτική αυτή στην πράξη έτσι ώστε οι τοπικές κοινωνίες να έχουν ένα αντιστάθμισμα και να μπορέσουν να αναπτυχθούν και να ζήσουν. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη και της εκπροσώπου από των ΗΕ προς την πρόταση αυτή. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Πριν δώσω το λόγο τον κύριο Williams, θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Ανίκη Γκαλάμα, συντονίστρια ε, από το ΒΒΕΦ. η οποία ε, έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό στο Κονγκό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να ασχοληθούμε με μια άλλη περιπτωσιολογική μελέτη και ελπίζουμε η κατάσταση να μην ε, εξελιχθεί με τον ίδιο τρόπο όπως στην Ιγυρία. Μιλώ για τον Εθνικό Δρυμό της Βαρούγκα, το παλαιότερο Εθνικό Δρυμό της Αφρικής, στην Ανατολική ε, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στα σύνορα με τη Ρουάντα και την Ουγκάντα. Αν το έχετε ακούσει, θα το έχετε ακούσει λόγω των ανταρτών που ζουν στις ορεινές περιοχές. Θα το έχετε ακούσει γιατί έχει εξαιρετικό φυσικό κάλος και εξαιρετική χλωρίδα και πανίδα, κυρίως τους γορίλες που ζουν σε πολύ ορεινά σημεία. Και βεβαίως βοηθιέται η τοπική κοινότητα. Σήμερα ο τριμός αυτός είναι γνωστός και για άλλο λόγο. Υποτίθεται ότι υπάρχουν πετρελαϊκά κοιτάσματα στην περιοχή. Η, η γαλλική Total και η αγγλικές εταιρείες έχουν μπει σε αυτό τον εθνικό δρυμό, σε αυτό το εθνικό πάρκο από το 2010 μέχρι και το 2011 και το 2012. Τους έχει παραχωρήσει τα εδάφη αυτά η κυβέρνηση του Κογκό για να ξεκινήσει η εκμετάλλευση. Όμως το 85% των υποτιθέμενων πηγών φυσικών πόρων και κοιτασμάτων είναι, βρίσκεται στον Εθνικό Πάρκο, στον Εθνικό Δρυμό, το οποίο έχει ενταχθεί στη Σύμβαση Ράμσαρ και ε, χέρι της προστασίας των Ηνωμένων Εθνών. Παρά τις ε, συγκρούσεις στο ανατολικό μέρος του Κονγκό, ε, το πάρκο έχει προστατευτεί αρκετά, είναι σε αρκετά σταθερή κατάσταση θα έλεγα σήμερα. Ταυτόχρονος, απαγορεύεται η αξιοποίηση των κοιτασμάτων βάσει διαφόρων διεθνών συμβάσεων μεταξύ των οποίων και συμβάσεις του ΟΗΕ. Μέχρι αυτή τη στιγμή καμία από τις ε, εταιρείες που ε, έχουν τις συμβάσεις παραγόρησης δεν έχει δηλώσει έχει δηλώσει ότι θα σεβαστεί την νομοθεσία και ότι θα τηρήσει αυτό που προβλέπεται, ότι απαγορεύεται δηλαδή αξιοποίηση και ανάπτυξη στην περιοχή. Η ΒΒΕΦ ανησυχεί ιδιαίτερως, χωρίς την πίεση από διεθνή φόρουμ, από διεθνή θεσμούς, τελικά θα αρχίσει η εκμετάλλευση αυτών των κοίτασμάτων και έτσι θα ε, τεθεί εν κινδύνο μια περιοχή μοναδική ε, στη γη, μοναδικού κάλους. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι ένα ζήτημα που μας ενδιαφέρει σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τη στιγμή που εμπλέκονται και ευρωπαϊκές εταιρείες Και βεβαίως ε, θα πρέπει σίγουρα οι ευρωπαϊκέ εταιρείε να εφαρμόζουν τους κανόνες της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της λογοδοσίας, εταιρικής λογοδοσίας, όταν δρουν και εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές του ε, και θα πρέπει οι κυβερνήσεις να μεριμνούν για την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών. Οι εταιρείε εγκατάλειψης πετρελαϊκών κοιτασμάτων και όταν λειτουργούν εκτός της επικράτειας ε, ε, θα, πρέπει να εφαρμόζουν τις ίδιες κατευθυντηρίες γραμμές. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Ανάπτυξη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει 30 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να βοηθήσει την ε, ε, κυβέρνηση του Κονγκό να ε, προστατεύσει τη βιοπικιλότητα και ένα τρίτο αυτών των κονδυλίων έχουν δεσμευτεί συγκεκριμένα για τη διατήρηση του Εθνικού Πάρκου του, της Βαρούνα. Μέχρι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει κάνει καλά πράγματα. Έχει κάνει μια πλήρη στρατηγική αξιολόγηση ε, περιβαλλοντική και έχει γίνει αξιολόγηση του αντικτύπου που θα έχει η αξιοποίηση πετρελαιοκών κοιτασμάτων στον εθνικό δρυμό εντός και ε, γύρω-γύρω από αυτόν. Θέλουμε να συμβάλλουμε στη διαδικασία και εμείς ε, ζητήσαμε από τις εταιρείε να σεβαστούν αυτή τη διαδικασία, να μην ξεκινήσουν δραστηριότητα πριν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, η οποία είναι ζωτική σημασία. Καμία από τις εταιρείε δεν έχει απαντήσει θετικά στο αίτημα αυτό μέχρι αυτή τη στιγμή. Αντιθέτως, έχουν ξεκινήσει τις δικές τους έρευνες. Ζητούμε λοιπόν από την Επιτροπή για την Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που έχει, να ασκήσει πίεση ούτως ώστε οι ευρωπαϊκές εταιρείες ε, να συμμορφωθούν με αυτή τη διαδικασία και να περιμένουν την ολοκλήρωσή της. Τελευταία παρατήρησή μου είναι η εξής. Θα ήταν εξαιρετικά θλιβερό το πετρέλαιο να αποτελέσει έναν ακόμα λόγο για οδύνη και ε, πόνο στη χώρα αυτή. Ελπίζουμε να μην αποτελέσει την επόμενη αιτία για σύγκρουση σε μια χώρα που έχει βιώσει εξαιρετικά πολλές ε, συγκρούσεις. Ε, το πετρέλαιο θα θέσει εν κινδύνο ένα μοναδικό μέρος στην Αφρική εάν τελικά επιτραπεί στις ε, εταιρείε να μπουν στο εθνικό αυτό πάρκο και να αξιοποιήσουν τα κοιτάσματα που υπάρχουν εκεί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις σας. Να δώσετε παρακαλώ την παρουσίασή σας και στη γραμματεία για να μοιραστεί σε όλα τα μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης. Τώρα κύριε Βουίλιαμς έχετε το λόγο. Θα σας προειδοποιήσω όταν εξαντληθεί ο χρόνος σας έχετε λίγη ώρα για να μπορέσει και η κυρία Κέμφ να απαντήσει στις ερωτήσεις Κορτές Λάστρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους όσους πήραν το λόγο. γιατί βλέπω ότι πολλοί από εσά παρακολουθούν την κατάσταση με ενδιαφέρον στην Ιγυρία. Και άκουσα και κάποιες προτάσεις οι οποίες έγιναν. Άκουσα και την παρατήρηση του κυρίου Ντίβα, δεν είναι εδώ πια. Μετά από την δολοφονία του Σαροντίουα, τα Ηνωμένα Έθνη, προσπαθεί με ένα, προσπαθούν με ένα πρόγραμμά του να εφαρμόσουν αυτά τα οποία ζητούσε ο Κέν κάποτε. Αγαπητά μέλη λοιπόν, σχετικά με αυτό το σκάνδαλο, και σχετικά με τις ε, αρμοδιότητες και τις εξουσίες ε, τις κρατικές, οι οποίες κανονικά δεν κάνουν αυτό που θα έπρεπε να κάνουν. Τα τελευταία χρόνια το λέμε αυτό συνεχώς στις εθνικές μας αρχές. Κάναμε ό,τι μπορούμε να πείσουμε ότι οι κρατικοί εταίροι πρέπει να λειτουργήσουν σωστά αλλά όλες οι προσπάθειές μας μέχρι τώρα απέτυχαν. Σχετικά με το flaring του φυσικού αερίου, τη διαδικασία αυτή, εγώ στράφηκα προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και στα πλαίσια της συνάντησης των εμπλεκομένων, των stakeholders, αναφερόμενος στις γνώσεις που έχουμε τις περιβαλλοντικές και μου ζητήθηκε να παρουσιάσω και την κατάσταση. Το έκανα αυτό, η πρότασή μου έγινε δεκτή από όλους τους εμπλεκομένους, αλλά δύο μήνες μετά ο τότε υπουργός ή ε, τότε υπουργός περιβάλλοντος εξεδιώχθη από τη θέση της. Και αυτή η πρόταση νομοθετική δυστυχώς απέτυχε. Πάντα οι πετρελαϊκές εταιρείες είναι αυτές οι οποίες επιβάλλουν την άποψή του και προφανώς στους νόμους μας υπάρχουν αυτά που είπατε για τις αδειοδοτήσεις. Εκεί όπου δεν ασκεί τη δραστηριότητα σύμφωνα με τη σύμβαση, ακόμα και στον τομέα του περιβάλλοντος, είχαμε ζητήσει ε, την εφαρμογή. Είχαμε πει ότι η Shell δεν είχε σεβαστεί τα επίπεδα τα οποία η ίδια είχε προτείνει αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει ισχύς από πλευράς των κυβερνήσεών μας, ούτε δεοντολογική, ούτε ηθική. Την ουσία, αν μας ζητάτε να κάνουμε ό,τι πρέπει, τότε θα σταματήσουμε την παραγωγή αν σταματήσουμε την παραγωγή δεν σας δίνουμε λεφτά για να μπορέσετε να ασκήσετε την κυβερνητική σας πολιτική. Λόγω λοιπόν αυτής της κατάστασης ε, έχουν χειροτερεύσει τα πράγματα. Δεν θέλουμε να ξεσπάσει η επανάσταση στην Ιγυρία, γιατί αν ξεσπάσει η επανάσταση θα είναι ένα πρόβλημα για το σύνολο του κόσμου. Αλλά έχουμε δυστυχώς φτάσει σε αυτή την άσχημη κατάσταση, συνειδητοποιούμε το τι συμβαίνει ακριβώς όπου υπάρχει και η Ισλαμική ομάδα Μπόκα Χαράμ που τρομοκρατεί και την κυβέρνηση και η κυβέρνηση δεν μπορεί καν να τους επαναφέρει στην τάξη. Αν η κατάσταση χειροτερεύσει περισσότερο τότε τα πράγματα θα είναι ανεξέλεκτα και γι' αυτό μια ευκαιρία που έχω να μιλάω μαζί σας και να θέτω τα θέματα είναι μια καλή ευκαιρία για μας. Σίγουρα οι κυβερνήσεις μπορούν να απειλήσουν για την αφαίρεση της αδειοδότησης, αλλά δεν θα το κάνουν, δεν τολμούν να το κάνουν. Και θα συμφωνήσω με την κυρία Κάλεμπ για τα διπλά στάνταρτ τα οποία επικρατούν. Προφανώς αυτά τα στάνταρτ που έχουν συμφωνηθεί έχουν συμφωνηθεί από όλους αλλά οι πολυεθνικές εταιρείες δεν σέβονται τις βασικές ε, συνθήκες τις οποίες εφαρμόζουν στις ε, πλούσιες χώρες, στις προχωρημένες χώρες. Οι μηχανισμοί επιβολής όμως στις χώρες αυτές είναι τέτοιοι που αναγκάζουν τις επιχειρήσεις να σεβαστούν ε, τις συνθήκες παραγωγής. Ενώ στις χώρες σαν τη δική μου, σαν την Ιγυρία, και υπήρξε επίσης και αναφορά και στην Δημοκρατία του Κονγκό, δεν έχει εκεί καταλήξει η κατάσταση. Και φοβάμαι ότι αν δεν αλλάξουν τα πράγματα στη χώρα αυτή, τότε θα μοιάσει αυτό που γίνεται στην Δημοκρατία του Κονγκό σε αυτό το οποίο γίνεται στην Ιγυρία και σε όλες τις άλλες χώρες όπου το πετρέλαιο είναι η βασική πηγή πλούτου. Η Γκάνα βέβαια προσπαθεί να δημιουργήσει μια εξαίρεση θα έλεγα σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες αφρικανικές χώρες. Γιατί εξ αρχής ε, πληροφορήθηκαν το τι γίνεται στις υπόλοιπες χώρες ε, και προετοιμάστηκαν εκ των προτέρων. Υπήρξε δηλαδή μια συνειδητοποίηση, μια κατάρτιση θα έλεγα, η οποία θα πρέπει να στηριχθεί και σε άλλες περιοχές όπως η Δημοκρατία του Κονγκό και το Σουδάν όπου το πετρέλαιο ε, ε, έχει αρχίσει να ε, διαφαίνεται σαν το βασικό στήριγμα της οικονομίας. Δύο επιπλέον ερωτήσεις έχουν τεθεί. Η πρώτη σχετικά με το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών. Και το λέω αυτό ξεκάθαρα. Χωρίς την κοινωνία των πολιτών ο υπόλοιπος κόσμος δεν θα είχε ιδέα για την κατάσταση στην Ιγυρία. Είναι δική μας ευθύνη όχι μόνο να μιλάμε σε αυτούς που είναι εκτός της χώρας, αλλά και σε αυτούς που είναι στις κοινότητες, στις χώρες μας. Η οργάνωσή μου ακριβώς είναι μια οργάνωση με βάση ε, λαϊκή και ενημερώνουμε τις κοινότητες ε, πώς θα προστατευθούν απέναντι στις καταστροφές που προκαλούνται από την πετρελαϊκή δραστηριότητα. Καταρχάς ζητάμε στις κοινότητες να μην εμπλακούν, γιατί κάποιες επιχειρήσεις πιστεύουν ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν και τα προβλήματα τα περιβαλλοντικά είναι, ε, προκαλούνται από το σαμποτάζ το οποίο ε, προκαλούν οι τοπικές κοινότητες. Αυτό μπορεί να έχει συμβεί μερικές φορές, αλλά στη μεγάλη περίπτωση των ατυχημάτων των οικολογικών ε, δεν οφείλεται σε σαμποτάζ κάποιων κοινοτήτων. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι το να λέμε ε, ότι οι περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις και τα ατυχήματα οφείλονται ε, σε παράνομες δραστηριότητες ή σε κλοπή γενικά δεν έχουν οι κοινότητες τους πόρους να ασκούν τέτοιες δραστηριότητες και πολλές φορές ε, τα στελέχη των επιχειρήσεων χρησιμοποιούν τις τοπικές κοινότητες για να κλέψουν ποσότητες καυσίμων. Απαιτείται λοιπόν πάρα πολύ προσπάθεια από πλευράς μας για να εκπαιδεύσουμε τους ε, κατοίκους των περιοχών, να τους συνειδητοποιήσουμε πολιτικά έτσι ώστε ε, κάποιες από τις ρυθμίσεις ε, να μην λειτουργούν αρνητικά. Και σαν δικηγόροι να προσπαθήσουμε μέσω του νόμου να πιέσουμε τις επιχειρήσεις να κάνουν αυτό το οποίο είναι σωστό. Αλλά δυστυχώς δεν ε, έχουμε αποτελέσματα επιθυμικά. Έχουμε αποφάσεις από τοπικά δικαστήρια, σαν παράδειγμα, εδώ και έξι χρόνια για να σταματήσει το φλέρινγκ του φυσικού αερίου αλλά η Shell συνεχίζει να το κάνει, να ασκολουθεί αυτή την πρακτική. Εγώ δεν έχω καθήκον και δυνατότητα να επιβάλλω τον νόμο. Ευθύνη μου είναι όμως είναι να πάω στα δικαστήρια, να τους ζητήσω να βγάλουν τις σωστές αποφάσεις και μετά είναι ευθύνη των κυβερνητικών αρμόδιων αρχών να θέσουν σε εφαρμογή τη συγκεκριμένη απόφαση. Σας ευχαριστώ λοιπόν και για τις ε, τελευταίες πρακτικές ε, ερωτήσεις τις οποίες κάνατε για το τι μπορεί να γίνει. Εμείς βλέπουμε τα πράγματα βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Το να αφήσουμε το πετρέλαιο ε, εκεί που βρίσκεται είναι μια τελευταία επιλογή. Εμείς με, αυτές, με αυτούς τους ελέγχους προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες μεσοπρόθεσμες προτάσεις. Έχουμε εμπλακεί άλλωστε σε, διεθνή, ε, σε, διεθνή, σε διεθνείς δικαστικές διαδικασίες, σε δικαστήρια της Χάγης εναντίον της ΣΕΛ. Αυτό είναι κάτι το οποίο θέτει ε, θέματα και νομικών δικαιοδοσιών γιατί θα πρέπει να υπάρχει δικαιοδοσία του δικαστηρίου να ασχοληθεί με τέτοια θέματα. Εν πάση περιπτώσει εμείς προσπαθούμε και θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα το επόμενο στάδιο. Αν χρειάζεστε τις δικές μου απόψεις για να, να κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις για την δυνατότητα χρήσης των δικαστικών δυνατοτήτων που υπάρχουν, γιατί όχι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά. Ως μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος συμφωνούμε όλοι ότι χρειαζόμαστε πληροφορίες για την κατάσταση. Αν είχατε την καλοσύνη να μας ενημερώσετε, να μας τηρείτε ενήμερους μάλλον, θα ήταν πολύ καλό. Τώρα θα σας ε, δώσω πάλι το λόγο κυρία Κέμπ. Μια και ακούστηκε μια ερώτηση που απευθύνονταν απευθεία σε εσά. Ναι, για να συνεχίσω και σας το είπε ο κύριος Βίλιαμ. Βεβαίως και η συνάδελφοι εδώ στις Βρυξέλλες ε, και εγώ ήμασταν πολύ ευτυχείς για την ε, εργασία μας στην ε, έκθεση της UNEP. Δεν νομίζω ότι επέκρινε την, έκθεση την ίδια ο κύριος Βίλιαμ, αλλά περισσότερο το γεγονό ότι δεν συμπεριελάμβανε τι ε, πετρελοκυλίδε τη τελευταία περίοδου στην ε, Ουγγουνιλάνδη. Ασφαλώ όμω παρακολουθούμε ιδιαίτερα τι δραστηριότητε εκεί τώρα στο Δέλτα του Νίγηρα. Και για την ερώτηση του κύριου Κορτές, ως προς τις ε, πρωτοβουλίες που υπάρχουν και που αναπτύσσονται ανά τον κόσμο ενδεχομένω ώστε να μην ε, υπάρχει αυτή η κατάχρηση των πόρων. Αυτή τη στιγμή η τάση είναι περισσότερο για την ε, διατήρηση της ε, κατάστασης όπως έχει. διαφύλαξη δηλαδή, της κατάστασης και όχι ε, φέρει από ψήλος των δασών για να προσφερθεί το προϊόν αυτής στους ε, ε, κατοίκους. Προσπαθούμε δηλαδή να τους κρατήσουμε στην περιοχή τους ταυτόχρονα με μια ε, δυνατότητα για ε, συμβίωση με τη φύση. Η διαδικασία είναι μακροχρόνια. Δεν μπορούμε να πούμε ότι μέσα σε ένα-δύο χρόνια μπορεί να γίνει τίποτα, αλλά από την άλλη πρέπει να σημειωθεί πρόοδο και βραχυπρόθεσμα για να μπορέσουμε να έχουμε προοπτικέ ανάπτυξη. Και βέβαια χρειάζονται μηχανισμοί παρακολούθησης, οι οποίοι θα αποτρέπουν τις ε, παραβιάσεις και που θα επιτρέπουν ταυτόχρονα την ε, συμμετοχή του πληθυσμού της περιοχής, ε, την παρακολούθηση από τον πληθυσμό της περιοχής της κατάστασης. Δεν θέλουμε δηλαδή εμείς επιθεώρηση αναγκαστικά άνωθεν, αλλά θέλουμε ουσιαστική διαφύλαξη της φύσης για το καλό των κατοίκων της περιοχής, όπως ε, άλλωστε αναφέρατε και εσείς στο Εκουαδόρ. Είναι ένα από τα, ε, ένας από τα προγράμματα ε, στόχους που έχουμε, μεταξύ άλλων, όπως το Βιετνάμ λοιπά. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Κέμφ Θα αφήσω το λόγο τώρα στην Σκακέλερ. Είχαμε πει ότι θέλαμε το χρόνο που έχουμε στη θέση μας να τον αξιοποιήσουμε για κάποια συμπεράσματα. Φυσικά. Ναι, ευχαριστώ, θα είμαι πολύ σύντομη. Ήταν πολύ σαφές νομίζω και πριν από τη δεξαγωγή βέβαια της ε, ακοράς ότι έχουμε σημαντική ε, επίδραση της ε, υποβάθμισης του περιβάλλοντος, της καταστροφής στην αποτυχία της προσπάθειας για της φτώχειας είναι κάτι το οποίο πρέπει όλοι να αντιμετωπίσουμε όπως και όλα τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπαθίες μας. Δεν προχωρούν στις αναπτυσσόμενες χώρες πράγματα που θα θέλαμε, αλλά πέραν αυτών μπορούμε νομίζω να κάνουμε κάτι και για την κλιματική αλλαγή ή για την προσφορά επαρκών πόρων για τις κυβερνήσεις εκείνες που θα τις βοηθήσει να προχωρήσουν στην ε, υιοθέτηση των μέτρων που χρειάζονται. Και επίσης πιστεύω ότι τα θέματα πρέπει να τεθούν επιτάπητος, πρέπει να προβλεφθούν στο πρόγραμμά μας και βέβαια θα πρέπει να δώσουμε και πολύ συγκεκριμένους ε, σαφείς στόχους και για το τι μπορούμε να κάνουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από πλευράς μας, αλλά και για το πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε άλλες χώρες. Η συμμετοχή της ε, τοπικής κοινωνίας των μη κυβερνητικών οργανώσεων είναι σαφώς, σαφές ότι χρειάζεται. Προβλήματα έχουμε όμως και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στο εσωτερικό δηλαδή ότι δεν, υπάρχουν, ε, δεν υπάρχει επαρκής ε, συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών σε σχέση με το περιβάλλον. Αυτό είναι ένα ακόμα έλλειμμα λοιπόν που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και εμείς από πλευρά μας, χωρίς να χρειάζεται να κατηγορούμε κανέναν άλλον. Πράσινη οικονομία έχει διαδραματίσει ρόλο φυσικά, πολύ σημαντικό. Δεν αρκεί όμως η οικονομία, χρειάζεται πολύ σημαντική ε, προσπάθεια. Και γι' αυτό καλό θα ήταν να βοηθήσουμε την οικονομία να προχωρήσει σε ανάληψη δράσης. από πλευρά τη, γιατί βέβαια θα πηγαίνει αυτή παράλληλα με τι επίσημε δράσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ θερμά. Γκάμπη, έχει το λόγο εσύ πάλι. Ευχαριστώ πολύ, Σκά. Ένα-δύο σημεία μόνο. Συμφωνώ ότι έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ευθύνη να κοιτάμε και το τι συμβαίνει στις ε, αναπτυσσόμενες χώρες να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή, να βοηθήσουμε στη διαφύλαξη της βιοπικιλότητας. Είναι πολύ σημαντικό να μην λησμονούμε ότι δεν υπάρχει μόνο η χρηματοπιστωτική κρίση ή η κρίση του ευρώ. Η περιβαλλοντική κρίση, οι στόχοι μας και η δέσμευσή μας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών της δεν μπορούν να ε, περισταλούν, δεν μπορούν να συμπιεστούν λόγω της οικονομικής κρίσης. και έτσι ενδιαφέρον άκουσα τις προτάσεις για, τα, ε, για τη χρήση της γης, για την ε, πτυτικότητα των ε, τιμών κτλ. Επίσης, θα πρέπει με πιο πολύ προσοχή να κοιτάξουμε το ρόλο των ευρωπαϊκών εταιριών στην υπόθεση αυτή. Δεν αρκεί νομίζω να μιλούμε για εταιρική ευθύνη. Πρέπει να κοιτάμε και την οικολογική ευθύνη και την ευθύνη για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε αναπτυσσόμενες χώρες και αυτό όχι μόνο με τις εθελοντικές δεσμεύσεις των εταιριών. Έχουμε διάφορους λόγους και τρόπους να μιλήσουμε για απευθείας ευθύνη για τις, ευθύν, για τις ζημιές που προξενεί η δράση αυτών των επιχειρήσεων και για συγκεκριμένες κυρώσεις. Δεν είναι δυνατό να περιοριστούμε ή να τις αφήσουμε ατιμόρυτες για τόσα έχουν πράξει. Και έτσι θα ήθελα να πω ότι σας στηρίζουμε στην, στον αγώνα σας για περισσότερη δικαιοσύνη, οικολογική και κοινωνική στις χώρες σας. Και βεβαίως θα παρακολουθούμε προσεκτικά όλες τις συζητήσεις. Ευχαριστώ όλους τους εδώ παριστομένους και κυρίως τον κύριο Williams όπως και την κυρία Κέμπ και ευχαριστώ θερμά και τους διερμηνείς για την παρουσία τους.